Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Κυρίσω την έναρξη της συνεδριάσεως της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Η ημερήσια διάταξη σας έχει αποσταλεί την 11η Ιανουαρίου Έχετε τυχόν σχόλιο όσον αφορά την λόγω ημερήσια διάταξη. Δεν νομίζω. Συνεπώς θεωρείται εγκεκριμένη. Έχω διάφορες ανακοινώσεις. Επρόκειτο να γίνει συνεδρίαση συντονιστών στις 5.30 ε, το απόγευμα σήμερα. Θα λάβει χώρα ανταυτού αύριο στις 11 και 4. Οπότε μπορείτε να περιμένετε εκτός της αιθούσης και όταν τελειώσει η συνεδρίαση θα ακούσετε τα πιο καινούργια νέα από τους συντονιστές. Θα το λέω για να το σημειώσετε ενδιαφερομένοι. Τα σημεία 10 και 11 τη ημερήσια διάταξη, απαλλαγή για του οργανισμού και απαλλαγή στι κοινέ επιχειρήσει κλπ. που ήταν για την 11η Ιανουαρίου, θα γίνει στι 24 Ιανουαρίου στι 3 το απόγευμα. Το 12 τη μέση διάταξη όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την απαλλαγή του είχε προγραμματιστεί για τις 3 αύριο το απόγευμα. Στις 5 θα γίνει η συζήτηση, αντί στις 3. Αυτά. Για αύριο σημείωστε διόντως, ενδιαφερόμενοι. Διατίθενται αρκετέ γλώσσες και τα πάντα εκπέμπονται και στο διαδίκτυο. Έχουμε νέο βοηθό στη γραμματεία, την κυρία Καρέλ Ντουλχώστ. Άκουσε πρόσδεκτη, καλώς ορίσατε, σηκωθείτε όρθια αν θέλετε να σας δούμε. Welcome. Καλώς ήρθατε. Στο σημείο 3 της ημερήσιας διάταξης πάμε στην εκλογή του Προεδρίου της Επιτροπής. Στο παράρτημα αναφέρονται ιδέες στις διαδικασίες. Σκοπός συνεδριάσεώς μας είναι η εκλογή ενός Προεδρίου πρέπει να εκλέξουμε πρώτα απ' όλα πρόεδρο και μετά αντιπροέδρους. Καταρχάς, πρέπει να διαπιστώσουμε ότι υπάρχει απαρτία το μεταξύ σας μέτρησα και είδα ότι πράγματι υπάρχει απαρτία. Υποψήφοι για τη θέση του Προέδρου μπορούν να προταθούν από τις πολιτικές ομάδες από τουλάχιστον 5% των μελών μπορούν να προταθούν. Είναι παλιά παράδοση ότι στα μισά της θητείας μπορούν να προταθούν νέοι υποψήφοι και θέλω να ρωτήσω αν οι ομάδες αισθάνονται την ανάγκη να προτείνουν κάποιον άλλον ε, ε, αντιπρόεδρο, κ. Χατζημαρκάκης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η ομάδα των Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη θα ήθελα να σας προτείνω Μιχαήλ Τόερε που είναι στα αριστερά μου εδώ και μέχρι στιγμής δεν ήταν μέλος της Επιτροπής μας αλλά έχει πολλή εμπειρία όσον αφορά τα δημοσιονομικά και τον έλεγχο του προπορισμού από τότε που ήταν ε, βουλευτής ε, στην τοπική βουλή της Βάδης ε, Βιδεβέργης. Μάλιστα με την κυρία Γκρέσλε διαχειρίζονται ένα προπορισμό πάνω από 40 δισεκατομμύρια ευρώ 14,5 έτη ήταν ε, δήμαρχος, ε, επικεφαλής δήμαρχος ε, στο Χόρτ, στη Βαντιβονιβόνη και εξελέγει με μεγάλο ποσοστό και θα χαιρόμουν να είχε παρόμοιο αποτέλεσμα και εδώ σήμερα. Εκτός μικροφώνου ο πρόεδρος. Michael. Ο Μάικλ. Α, δεν υπάρχει άλλος υποψήφιος. Άρα ο κύριος Μάικλ Τόρερ είναι ο νέος πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου του Προπολογισμού. Του εύχομαι κάθε επιτυχία στη νέα αυτή σημαντική του θέση. Παρακαλώ, ελάτε να πάρετε τη θέση μου. hello. Uh, Γεια σας, ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποστήριξή σας. Είναι τιμή μου που είμαι εδώ. Έχω ήδη κάποιες, κάποιους που θέλουν να πάρουν το λόγο. Uh, Ως πρόεδρος της ε, Επιτροπής αυτής θα περάσω τώρα στην ε, γλώσσα τη μετρική μου. Η κυρία Ίγκεμπορ Κρέσλα έχει πρώτη ζητήσει το λόγο. Ξενόμως στο ΕΛΚ, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σα ε, ευχαριστήσω τον κύριο Μουλή για την πολύ καλή εργασία του. Μια που οι φιλελεύθεροι για πρώτη φορά στον ομάδα αυτό επέτρεψαν να έχουν ένα πρόεδρο της Επιτροπής που ξέρει τα πράγματα και έχει εμπειρία. Θα ήθελα να εκφράσω την ε, τις προσδοκίες που έχει αυτή η Επιτροπή και η μεγαλύτερη πολιτική ομάδα ότι θα ήταν ωραίο που να εκλέγαμε ένα ενεργό μέλος. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα σας, δεν θα σας ε, καλοδεχθούμε, αλλά θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Μούλτερ, γιατί η Προεδρία ήταν σε πολύ καλά χέρια όσο ήταν εκείνο πρόεδρος και να πω ότι πραγματικά ε, απολαύσαμε την Προεδρία του να είναι πρόεδρος, δηλαδή κάποιος ο οποίος ξέρει τα πράγματα τόσο καλά και ιδίως τα θέματα της Επιτροπής Ελέγχου του Υπουργορισμού. Σε ευχαριστώ Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ. Σα ναι, σας ευχαριστώ κύριε Κρέσλε. Τα πολλά χειροκροτήματα δείχνουν ότι η Επιτροπή ευχαριστεί πραγματικά τον πρόεδρο Γιάνν Μούλτερ για την εργασία του. Ο κύριος Γκάιαρ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να σας ευχηθώ κάθε επιτυχία στο αξίωμά σας. Είναι πολύ καλό αυτό το έργο που αναλαμβάνετε, αλλά δεν είναι πάντα εύκολο. Γιατί η Επιτροπή αυτή πολλές φορές είναι πολύ ιδιάζουσα. Ε, εξετάζουμε όλους τους τομείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολλές φορές ε, οι εργασίε μας δεν μας κάνουν και πολύ αγαπητούς στους συναδέλφους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γιατί πολλές φορές δεν ασχολούμεθα μόνο με τον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου και καμιά φορά αναγκαζόμαστε να συζητήσουμε με κάποιους συναδέλφους και το πώ είναι λογικό κάτι που έχουν προτείνει και έχουμε οκρές συζητήσει από αυτόν ταυτόχρονα όμω, εξετάζουμε την πολιτική του Προεδρείου του Σώματος και ελέγχουμε τις αποφάσεις που λαμβάνονται εκεί όσον αφορά την εκτέλεση του προπολισμού. Θα το συστήσουμε κατά τη συνεδρία αυτή με στα πλαίσια της ε, απαλλαγής. Καταρχήν λοιπόν θα ήθελα να σας ευχηθώ κάθε επιτυχία στο αξίωμά σας και εγώ προσωπικά θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Γιάν Μούλτερ και εξ της πολιτικής μου ομάδας. Πολύ καλά εργάστηκες Γιάν. και θεωρώ ότι πραγματικά ήταν παραδειγματικό ο τρόπος με τον οποίο προέδρευσε στον εργασιών μας. Ε, Τα πρόχνω να πω ότι πήρα το λόγο για να πω ότι θα πρέπει τώρα βέβαια να περάσουμε στην εκλογή των αντιπροέδρων. Είναι σωστό ότι ο πρώτος αντιπρόεδρος της Επιτροπής αυτής, μια που ισχύει ε, ο κανόνας Ντόντο, είναι ε, από τους σοσιαλδημοκράτες και συζητήσαμε την υποψηφιότητα της κυρίας Αντρεάσεν και θα σας πούμε γιατί εμείς δεν υποστηρίζουμε την υποψηφιότητα της Μάρτη Αντρεάσεν. Θα θυμούνται οι συνάδελφοι ίσως. Νομίζω ότι αυτό έγινε κατά τη διάρκεια της συζήτησης απαλλαγής ε, του προπολισμού του Κοινοβουλίου πέρσι, όπου είχαμε μια κατάσταση κατά την οποία, αν δεν κάνω λάθος, η Daily Mirror ή μια παρόμοια βρετανική εφημερίδα υψηλής ποιότητας δημοσίευσε κάποιο αριθμητικό στοιχείο ε, του οποίου η πηγή ήταν η κυρία Αντρέασεν. Δηλαδή ότι το αναμενόμενο κόστος ε, του οίκου για την ευρωπαϊκή ιστορία ήταν, αν θυμάμαι καλά, 120 με 150 εκατομμύρια. Τότε στη συζήτηση είχα ρωτήσει ποια ήταν η πηγή, γιατί είναι πολύ περίεργο αυτό. Να υπάρχει δηλαδή κάποιος αριθμός για τον οποίο εκτός από μια βουλευτή που θεώρησε ότι είναι λογικό αυτό το αριθμό δεν υπήρχαν άλλες πηγές. Ούτε η εφημερίδα, ούτε η κυρία Αντριάσεν, μέχρι σήμερα δεν ε, έκανε δώσαν καμία εξήγηση γι' αυτό. Και ομολογώ ότι αυτό ούτε κοινοβουλευτικά μου φαίνεται πολύ επικοδομητικό, ούτε πολύ σοβαρό. Λόγω αυτού η δική μου πολιτική ομάδα δεν προτίθεται να υποστηρίξει την υποψηφιότητα της κυρίας Αντρεάσεν. Πρώτος αντιπρόεδρος ήταν ο κύριος Στάς μέχρι στιγμής των Πρασίνων. Νομίζω ότι εργάστηκε πάρα πολύ καλά και αν δέχεται να συνεχίσει το έργο του έχει την απόλυτη υποστήριξή μας. σε ευχαριστώ κύριε Γκάιε. Από ό,τι κατάλαβα είμαστε τώρα στο σημείο εκλογή των αντιπροέδρων όπου υπάρχει συζήτηση. Ξεκίνησε η συζήτηση για τα πρόσωπα που προτείνονται όσον αφορά την πρόταση της ΕΦΤΕ που έχει το δικαίωμα σύμφωνα με το ε, όντα. Υπάρχει κάποιος από την ομάδα CFT που θέλει το λόγο. Φαίνεται όχι. Α, ναι. Äh, Με ενημερώνουν ότι ο Στάνφος Έγνου θέλει το λόγο. Yes, good afternoon. I am substituting. Καλησπέρα. Αντικαθιστώ τον Μάριν Είμαι ονομά Άγνιου. Είμαι από την ομάδα EFT βάσει των όσων υπόθηκαν. Δηλαδή ότι η δημοσιογράφος έκανε το σφάλμα και όχι η κυρία Ανδρίασον. Αυτό ήθελα να πω. Okay. Ναι, Άρα. Τώρα αυτό δεν ε, σχετίζεται βέβαια με το συγκεκριμένο ε, άτομα. Θα ήθελα να παρακλέσω τον άδελφο Γιάνν Μούλτερ, ο οποίος έχει ενημερωθεί ότι η συνάδελφος δεν μπορεί να είναι παρούσα σήμερα αληθεύει ότι σας έστειλε μία αποστο... επιστολή ότι βρίσκεται στο νοσοκομείο σήμερα, κύριε Μούλτερ, μπορείτε να μας πει κάτι από αυτού. Ναι. Νομίζω την περασμένη εβδομάδα, Τετάρτη, Πέμπτη, δεν είμαι σίγουρος, ήρθε στην Ολομέλεια και μου έδωσε μία επιστολή που απευθυνόταν προς τον πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου Προεπολογισμού... και ανέφερε στην επιστολή ότι είναι υποψήφια. Παρέδωσα την επιστολή στην ε, γραμματεία στο Στρασβούργο και την Πέμπτη όταν επρόκειτο να φύγω το απόγευμα είπα να στείλει ηλεκτρονικό μήνυμα στη γραμματεία και δια της ηλεκτρονικής οδού. Νομίζω ότι με τρεις τρόπους ε, ενημερωθήκαμε ότι είναι υποψήφια. Δεν μπορούσε να παρίσταται διότι έπρεπε να παραστεί σε μια ε, συνάντηση που δεν μπορούσε να βάλει πλέον. Ευχαριστώ πολύ, λέει από ό,τι μας λέγουν είναι υποψήφια και πρότεινε ο συνάδελφος Γκάιερ και άλλον υποψήφιο και θα λάβει χώρα ψηφοφορία αλλά ζήτησα πρώτα απ' όλα να μου πείτε κατά πόσον ε, θέλει κάποιος να μιλήσει. Ο κύριος Χατζημαρκάκης. Καταρχήν, Πρόεδρε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και εξ των συστικής πολιτικής ομάδας κάθε επιτυχία. Η συνάδελφο Γκρέσλε αναφέρθηκε ότι θα πρέπει να βασιζόμαστε στην εμπειρία πολλέ φορέ. Το κάναμε αυτό και είμαστε πολύ υπερήφανοι για την εργασία του Γιάνν Μούλτερ, όχι μόνο στο εξάμεινο που ήταν πρόεδρο, αλλά καθ' όλη τη διάρκεια τη θητεία του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί είναι πραγματικά από του γνώστε, του πιο ικανού γνώστε των θεμάτων. Και αυτό η ομάδα μου είναι ιδιαίτερα ευγνώμων για την εργασία του. Όσον αφορά τώρα την υποψιότητα του ε, κυρίας Αντρέασεν, το σχόλιο της ε, κυρίας Γκρέσλε προς συναδέλφους ε, είναι σχετικό γιατί σχετίζεται με το σύστημα DONT. Ω εκπρόσωπο μια πολιτική ομάδα που προ το παρόν δεν είναι τόσο μεγάλη, θέλουμε να τηρούνται οι κανόνε DONT. Το θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και γι' αυτό, στον πρώτο γύρο, θα θέλαμε να παραμείνει αυτή η συμφωνία που έχει υιοθετηθεί από το Κοινοβούλιο. Εάν δεν έχει επαρκούς ψήφους η κυρία Αντρέασεν, ευχαρίστως να ε, ξανακαλωσορίσουμε τον Σνάλφο Μπαρτστάς στο Προεδρείο, γιατί όχι μόνο συνεργαστήκαμε πολύ καλά μαζί του, αλλά κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους πολλές φορές ανέλαβε το θόκο του Προέδρου και πραγματικά ήταν πάρα πολύ ικανός πρόβλημα. Λοιπόν, θα μπορούσαμε κάλλιστα να υποστηρίξουμε των Στάς, ε, Είναι η πρόταση των σοσιαλδημοκρατών. Πρόεδρος. Ωραία, θα πρέπει να διευκρινίσουμε τώρα τη διαδικασία. Πριν ε, υποβάλω μια ερώτηση προς τον Στάτ, ο κύριο Γκάιαρ έχει στήσει το λόγο. Εγώ θα ήθελα να αντιδράσω σε αυτά που είπε ο κ. Άγνιο. Γιατί αν έχει δίκιο θα μπορούσαμε να αξιολογήσουμε διαφορετικά τη διαδικασία, αλλά εγώ το θυμάμαι τελείω διαφορετικό. Γιατί κατά τη διάρκεια τη συζήτηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο ε, παρακάλεσα από την κυρία Αντρεάς να διαθέσει τα στοιχεία αυτά στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Γιατί βέβαια θα θέλαμε να ελέγξουμε τις πηγές των στοιχείων αυτών, γιατί είναι πολύ ε, αφισβητούμενο ε, θέμα ο οίκος της Ευρωπαϊκής Ιστορίας. Και βέβαια το κόστος είναι κάτι που ενδιαφέρει τις Επιτροπές Προϋπολογισμού και Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Και μέχρι στιγμής δεν είχαμε καμία αντίδραση από την κυρία Αντρεάσεν. Γι' αυτό υπέβαλα την πρόταση που υπέβαλα. Πρόεδρος. Ωραία. Η πρόταση είναι να μην κάνουμε εδώ συζήτηση ε, επί προσώπων, ιδίω μια που η εν λόγω δεν μπορεί να είναι παρούσα. Γι' αυτό θα θέλαμε να περάσουμε στην ψηφοφορία. Προτείνονται δύο υποψήφοι. Από τη μία ξέρουμε γραπτά ότι είναι διαθέσιμη. Ε, προτάθη επίσης ο Μπαρτ Θα θέλω να ρωτήσω τον κύριο Στάς είναι υποψήφιο πραγματικά στον πρώτο γύρο. Αυτή νομίζω είναι η σωστή διαδικασία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Την προηγούμενη φορά είχε υπάρξει πρόταση από τη διάσκεψη των Πρόεδρων για την εφαρμογή του κανόνα ΔΕΟΝΤ. Η κυρία Αντρέασεν ήταν υποψήφια την οποία πρότεινε η ομάδα EFT. Ω μέλο μια ε, μικρή ε, πολιτική ομάδα συμφωνώ με τον κύριο Χατζημαρκάκη, που βέβαια δεν εκπροσωπεί μια μικρή, αλλά μια μεσαία, μεσαίου μεγέθους ομάδα. Νομίζω όμω ότι για όλε τι μικρομεσαίε ομάδες καταρχά θα πρέπει να εφαρμοστεί ο κανόνα DON'T. Επομένως, η διαδικασία θα ήταν η εξή. Να δούμε αν στην Επιτροπή μα υπάρχει αρκετή υποστήριξη ώστε καταρχά να ακολουθηθεί ο κανόνα διόν που πρότεινε η διάσκεψη των Προέδρων και εν συνεχεία ίσω θα μπορούσαμε να έχουμε ένα δεύτερο γύρο με άλλου υποψηφίου εάν δεν ε, υπάρξει αρκετή υποστήριξη εδώ στην Επιτροπή μα ε, για την εφαρμογή του κανόνα Ντεόντ. Εγώ πάντως εφόσον ε, προκύψει αυτό, δέχομαι ε, να υποβάλω υποψηφιότητα και εγώ. Άλλωστε, νομίζω ο κύριος Αντρέασεν με είχε προτείνει ως υποψήφιο την προηγούμενη φορά, παρότι τελικά δεν είχε ε, γίνει δεκτή. δεν, ξέρω ακριβώ τι είχε γίνει τότε. Ο κύριο και οι σοσιαλιστές από ό,τι φαίνεται με στηρίζουν. Εάν ισχύει αυτό, ναι, μπορώ ευχαρίστως να σας πω ότι θα είμαι υποψήφιος. Ωραία, σας ευχαριστώ. Διευκρινίσουμε λοιπόν την κατάσταση. Μπορούμε να ακολουθήσουμε αυτή την άγουσα. Η πρόταση της διάσκεψης των Πρόεδρων υπάρχει, βάσει της οποίας ε, προτείνει η κυρία Αντριάσεν. Θα περάσουμε στην ψηφοφορία και ανάλογα με το αποτέλεσμα θα δούμε κατά πόσο θα χρειαστούμε και μια άλλη λύση ή όχι. Δεν βλέπω να διαφωνεί κανεί, Λοιπόν, θα ψηφίσουμε. Το είναι η Μάρτια Ανδρεάσεν. Και θα πρέπει η ψηφοφορία αυτή να γίνει γραπτά. Παρακαλώ να μοιράσετε τα ψηφοδέλτια. Äh, äh, θα πρέπει να έχουμε κάποιου ψηφολέκτε. Νομίζω θα πρέπει όλε οι πολιτικέ ομάδε να συμμετάσχουν στη δικασία αυτή. Äh, Υπάρχουν ε, θελοντές, η Ευρωπαϊκή τώρα θέλει λόγω των μελλοντικών του καθηκόντων από του σοσιαλιστέ, υπάρχει κάποιος που θέλει να είναι ψηφολέκτης, προτείνεται κάποιον. Frau Kollegin Prosperata oder Kollege Safrakakis. Προσπεράτα, ωραία. Ρόφος Χατζημαρκάκης. Άλλος που θέλει να καταμετρήσει. Αρκούν, αρκούν, ωραία. Μπορούμε να ξεκινήσουμε λοιπόν. Παρακαλώ να μοιραστούν τα ψηφοδέλτια αυτή τη στιγμή. Έχουμε 20 μέλη της Επιτροπής μας παρόντα. Παρακαλώ να μοιράσετε τα ψηφοδέλτια. Okay, die Stimmzettel werden jetzt an die anwesenden Mitglieder. Λοιπόν, διανύμονται τα ψηφοδέλτια στους παρόντες ε, βουλευτές που είναι μέλη της ομάδας αυτής, της ε, επιτροπής αυτής και μπορέσουμε μετά να ψηφίσουμε. Gibt es Rückfragen noch? Ερωτήσεις? Δηλαδή στο ψηφοδέλτιο θα βάλουμε ναι ή όχι, τι, θα, τι πρέπει να κάνουμε δηλαδή. Πρόεδρος, όταν μοιραστούν τα ψηφοδέλτια θα σας δώσω τις απαραίτητες οδηγίες. so das sekretariat hat mich Λοιπόν, δεν είναι προετοιμασμένα τα ψηφοδέλτια. Θα υπάρχουν με ναι ή όχι ή με αποχή. Και θα σα καλέσω ονομαστικά να παραδώσετε τα ψηφοδέλτια σα. Σε λίγα λεπτά θα υπάρχουν τα ψηφοδέλτια αυτά. Δεν είναι ακόμα έτοιμα. Okay. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, μοιράζω τώρα τα ψηφοδέλτια. Προτινόμενη υποψήφιο είναι η Μάρτα Ανδρεάσεν. Έχετε τη δυνατότητα να ψηφίσετε ή ναι ή όχι. Και αν δεν ψηφίσετε ούτε ναι ούτε όχι, θα θεωρηθεί ότι έχει πρακτική αποχή. Και θα πρέπει να δούμε ποια θα είναι ε, η πλειοψηφία των ε, ψήφων. Θα καλέσω τους αδέλφους εδώ για να παραδώσουν την ψήφο σας. Κύριε Ήταλε, θέλετε να έρθετε να είστε και εσείς εδώ, μια που είστε ψηφολέκτης. Λοιπόν, έχουν όλοι το ψηφοδέλτιο. Λοιπόν, άρχεται η ψηφοφορία. Θα σας καλέσω ονομαστικά.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 Επόμενος Ντορικ Βόλ. Der nächste ist Bojoslav Liberatsky.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 The next is Theodoros Skylakakis. is Yorgos Stavrakakis. Und dann Sören Bo Söndergaard.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 Paul Rübig. Kollege Czarnecki. Und Michael Theurer.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 Uh, Υπάρχει κάποιο συνέδριος που δεν έχει ψηφίσει ακόμα. Όχι. Ωραία. Ολοκληρώνεται η ψηφοφορία. Παρακαλώ τους ψηφολέξει να καταμετρήσουν. Α, όχι κι άλλο ένα συνέδριο. Χάρτο, γι' συνάδελφος. Χάρτογκ. Γι' αυτό ρώτησα, κύριε Χάρτογκ. Παρακαλώ. Έχετε το δικαίωμα ψήφου. Παρακαλώ. Λοιπόν, ολοκληρώνεται εδώ οριστικά η ψηφοφορία. Liebe Kolleginnen Kollegen. Αγαπητοί συνάδελφοι, περνάμε στην μεσαία διάταξη πάλι. Μετά την καταμέτρηση των ψήφων έχουμε το εξή αποτέλεσμα. 22 παρόντες ε, βουλευτέ με δικαίωμα ψήφου, μία αποχή, 10 μέλη έχουν ψηφίσει ναι και 11 όχι. Άρα η υποψήφιος δεν επέτυχε την απαραίτητη πλειοψηφία. Και περνάμε λοιπόν σε ένα δεύτερο γύρο. Ένα δεύτερο γύρο όπου από την προηγούμενη συζήτηση είδαμε ότι υπάρχει κάποιος υποψήφιος. Υποθέτω ότι παραμένει η πρόταση του αδέλφου Γκάιερ επιτάπητος. Άρα, ξαναρωτάω τώρα τυπικά το κύριο Στάς κατά πόσο είναι υποψηφί στο δεύτερο αυτό γερό. Ναι, δέχομαι ε, να είμαι υποψήφιος. Er λοιπόν, ο κύριο Στάση είπε ότι συμφωνεί. Äh, äh, Και μου είπανε ότι οι υποψήφοι πρέπει να δηλώσουν κατά πόσον έχουν συμπληρώσει τη δήλωση για τα οικονομικά του συμφέροντα. Νομίζω ότι έχει γίνει αυτό. Μάλιστα. Ωραία. Μπορούμε σε ένα δεύτερο γύρο να ψηφίσουμε τώρα. Gibt es hier Wortmeldungen? Wie das? Θέλει κάποιο το λόγο? Äh, λοιπόν, ένα συνάδελφο ε, ρωτάει τι θα γίνει εάν όλοι συμφωνούν. Στην περίπτωση δεν χρειαζόμαστε ένα δεύτερο γύρο, αλλά δεν νομίζω. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε τυπική ψηφοφορία. Γιατί με το, λόγω τη αποσύρσης τη κυρία Αντρεάσεν ε, δεν μπορεί να αποσύρει την ψηφοφορία τη. και γι' αυτό θα ήθελα να σα να σας συστήσω να είμαστε σίγουροι και να κάνουμε ένα γύρο ψηφοφορίας με δύο υποψηφίους. Επί η κυρία Γκρέσλε. Μα δεν κατάλαβα. Γιατί παραμένει η κυρία Αντρεάσεν στο ψηφοδέλτιο. Δεν το καταλαβαίνω. Warum Γιατί όχι, λέει ο πρόεδρος. Κοιτάξτε, μια που δεν είναι παρούσα, δεν μπορεί να αποσύρει κανένα την ψηφοφορία τη. Sie müsste neu vorgeschlagen Μα έχει προταθεί γραπτά από την ομάδα τη. Και γι' αυτό λέω ότι θα πρέπει να κάνουμε ε, μια ψηφοφορία με τους δύο υποψηφίους. Αλλά εάν το βλέπετε διαφορετικό, παρακαλώ, να έχουμε μια σύντομη συζήτηση. Ο κύριος Χατζημαρκάκης. Μα έχει δίκιο ο πρόεδρος. Μια που δεν έχουμε τη σύμφωνη γνώμη της ότι δεν είναι υποψήφια, παραμένει υποψηφιότητά της. Εκτός αν η ομάδα της αποσύρει την υποψηφιότητα. Αλλιώς πρέπει να ψηφίσουμε. Äh, Ευχαριστώ. Προφορικά μου είχε πει η κυρία Αντρέασον ότι εάν δεν γίνει δεκτή υποψηφιότητά τη, στο δεύτερο γύρο θα στηρίξει τον κύριο Στάς. Ε, Α, ναι, αν έχουν έτσι τα πράγματα. Θεωρούμε δηλαδή ότι αποσύρει την υποψηφιότητά τη για το δεύτερο γύρο. Άρα έχουμε ένα μόνο υποψήφιο, τον Μπαρτ Στάς. Άλλες υποψηφιότητες για την πρώτη ανυπροεδρία της ε, Επιτροπής μας. Όχι. Μπορούμε δηλαδή διαβοήσει να ψηφίσουμε τον κύριο Στάς. Συγχαρητήρια κύριε Στάς. Λοιπόν, περνάμε στην εκλογή του Δευτέρου Αντιπροέδρου. Προτάσεις παρακαλώ. Who is who is proposed yes. for the second? Yeah. yeah. hmm? Gressle hat das Wort. Ja, ich möchte. Kira Γκρέσλε, για το ΕΛΚ θέλω να προτείνω τον συνάδελφο Ζώνη από την Πολωνία. Ζώνιχ ε, είναι εδώ. Όχι, συγγνώμη, κάτι μπέρδεψα, λέει η κυρία Γκρέσλε τη συνάδελφο Ιβάνοβα από τη Βουλγαρία ήθελα να προτείνω, έκανα λάθος. Λοιπόν, δεν έχουμε δηλαδή δύο υποψήφιου, μία υποψήφια μόνο, την κυρία Ιβάνοβα. Άλλε προτάσει. Όχι. Ωραία. Αν συμφωνείτε, μπορούμε και εδώ διαβοή να ψηφίσουμε. Συγχαρητήρια, κυρία Ιβάνοβα. Ελπίζω να συνεργαστούμε πολύ ωραία. So, dann στον τρίτο αντιπρόεδρο. Πράγει κυρία Κρέσλε, έχει το λόγο. Ναι, ναι, αυτό εννοούσα προηγουμένω, το Σάλβο Σόνικ. Ωραία. Αυτό είναι όμω ο υποψήφιο για την τέταρτη αντιπροεδρία, νομίζω. Υπάρχει πλήρη σύγχυση. Γιατί για τον τρίτο αντιπρόεδρο είναι ο Ούσαφ Φολάτσκι από του Σοσιαλιστέ ε, για να παραμείνουμε στη δικασία. Ja, die Kollegin ist ο συνάδελφος Λιμπράτσκι προτείνεται, είναι πίσω σα, ναι, ναι, σωστά. Άλλη πρόταση, όχι, λοιπόν, εξελέγει ο συνάδελφος Λιμπράτσκι, συγχαρητήρια. Λοιπόν, η κυρία Γκρέση λέει, με συγχωρείτε, ζητώ συγγνώμη τον κύριο Σόνικα, αλλά έτσι και εγώ σήμερα μόλις τον γνώρισα. Λοιπόν, ο κύριο Σόνικα από την Πολωνία προτείνεται για τέταρτη προεδρία. Ευχαριστώ, λέει πρόεδρο. Άλλε προτάσει όχι. Μπορούμε και εδώ διαβοή λοιπόν να τον εκλέξουμε. Συγχαρητήρια κύριε Σόνικ. Ελπίζω να συνεργαστούμε πολύ ωραία. So, vielen Dank. Damit haben wir die Ευχαριστώ. Ολοκληρώθηκαν λοιπόν εδώ οι ψηφοφορίε. Επιτυχώ. Στη δημοκρατία καμιά φορά βέβαια αυτό κοστίζει κάποιο χρόνο. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Und können dann zum nächsten Tagesordnungspunkt äh, kommen. Μπορούμε να γράψουμε στο επόμενο σημείο τη ημερησία διάταξη. Έγκριση των πρακτικών τη συνεδρια 29 Νοεμβρίου και 8 ε, Δεκεμβρίου 2011. Παρατηρήσει από αυτόν, από ό,τι φαίνεται όχι. Εγκρίνονται λοιπόν και μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο σημείο, σημείο 5 τη ημερήσιας διάταξη. Απαλλαγή 2010, Γενικός Προπολογισμό τη Ευρωπαϊκής Ένωση. Θα θέλαμε εδώ να καλωσορίσουμε καλύτερα την Επίτροπο, που νομίζω τώρα έρχεται. Α, Καλώς ορίσατε κυρία Πέτρο και Κουίν. Με συγχωρείτε για την καθυστέρηση, αλλά είδα η της Δημοκρατία οι εκλογέ που είχαμε να κάνουμε. Λοιπόν, τώρα θα ήθελα καταρχήν να δώσω το λόγο στον ή μάλλον να χαιρετήσω τον υπεύθυνο ηλεκτρικού συνεδρίου, τον κύριο Λάτισλαβ Μπάλκο. να κάνετε μια εισαγωγή. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Καταρχά δράτω με τη ευκαιρία για να σα συγχαρώ για την εκλογή σα στη θέση του Πρόεδρου τη σημαντική αυτή επιτροπή. Συγητή κ. Φιόλνερ, αγαπητέ κύριε Συγητά, κ. Φιόλνερ, αγαπητά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να χρησιμοποιήσω αυτή την ευκαιρία στα πλαίσια δικασία απαλλαγή για το οικονομικό έτος 2010 να σα ενημερώσω συντομία για την προσέγγιση που ακολούθησε το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο όσον αφορά τον έλεγχο χρηματοδοτήσεων προγραμμάτων για την έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη που είναι σημαντικό σημείο των δαπανών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και αυτά αναφέρονται στο κεφάλαιο 6 της ετησίας εκθέσεως του ελεγκτικού συνεδρίου. Σαν συνεισηγητής για τον έλεγχο του τομέα θα ήθελα να δηλώσω όσον αφορά την σύνθεση του κεφαλαίου 6 ότι είναι νέο κεφάλαιο της ετήσιας εκθέσεως. Ε, δηλαδή ένα τμήμα αυτού το 2009, στην έκθεση του 2009 ήταν στα κεφάλαια 5 για έρευνα, ενέργεια και μεταφορά, 7 για παιδεία και ηθαγένεια και κεφάλαιο 8 οικονομικές και χρηματοπιστωτικές υποθέσεις. Αυτό εξηγείται και στην παράγραφο 1.10 της ετήσιας έκθεσης, όπως θα σας ενημέρωσε η συνάδελφός μου η κυρία Κέλουλάιτ στη συζήτηση που έγινε από το κεφαλαίο 1, εδώ σε αυτή την Επιτροπή αρχές Δεκεμβρίου. Ένας βασικός λόγος για τους οποίους το ελεκτικό συνέδριο επαναμοδοποίησε τον έλεγχο τι ομάδε πολιτική των έλεγχο είναι διότι ήθελε πιο αποτελεσματική ανάλυση των δαπανών τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω, λαμβάνοντα υπόψη τους κινδύνους που αντιπροσωπεύουν οι διάφοροι τομείς πολιτικής. Παρόλο που το ποσοστό σφάλματος στα πλαίσια του παλαιού κεφάλαιου 5 για την ενέργεια μεταφορές και το 6 έρευνες και εσωτερική πολιτικής δεν μπορεί να συγκριθεί άμεσα, δεν μπορεί να συγκριθούν μεταξύ του άμεσα, αλλά παραμένουν κάποιε σημαντικέ ομοιότητε. Πρώτα απ' όλα και στι δύο περιπτώσει οι περισσότερε ψυχικέ διαπάνε για τι διάφορε ομάδε πολιτικών αποτελείται από την έρευνα για τα προγράμματα. Ήταν περίπου 70% στο πρώτο κεφάλαιο 5 και 63% στο παρόν κεφάλαιο 6. Ε, Δεύτερον, 2% ήταν το, σφάλμα, ε, ε, το επίπεδο σφάλματο στο κεφάλαιο 5 και είναι ακόμα 4% στο κεφάλαιο 6 το 2010. Βασικός, βασική πηγή σφαλμάτων το 2009 και το 2010 ήταν ίδια. Επιστροφές μη επιλέξιμων ή ανακριβώ δηλωθέντων δαπανών για έρευνα των διαφόρων ε, προγραμμάτων και τι ενδιάμεσε πληρωμέ. κάτι που διαπίστωσε ε, και το 2010 ότι υπήρχαν σημαντικά σφάλματα και συχνά γινόταν. Τα πορίσματά μας εστιάζονται στις πληρωμές όσον αφορά την ερευνητική πολιτική στα κεφάλαια μάλλον στο 6ο και 7ο πολιτέ πρόγραμμα πλαίσιο. Εκεί υπάρχουν πολλαπλά προγράμματα που υποστηρίζουν διάφορου θεματικού τομεί και διάφορα είδη προγραμμάτων. Βασικό χαρακτηριστικό των προγραμμάτων είναι και το εξή. Εφαρμόζονται κατά βάση υπό άμεση κεντρική διαχείριση η εξολόγηση του κινδύνου για τα ασθαλείς είναι εξή, ότι οι δικαιούχοι ίσως συμπεριλαμβάνουν αδικαιολόγητες δαπάνες τους αξιώσεις τους, που να μην διορθώνονται από τους εποπτικούς φορείς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πριν επιστραφούν τα χρήματα. Αυτός ο κίνδυνος ενισχύεται από την περιπλοκότητα των κανόνων για τον υπολογισμό των επιλεξιμών δαπανών και την απέτηση οι δικαιούχοι να κάνουν σωστού υπολογισμού και να μην συμπεριλαμβάνουν μια επιλέξιμα στοιχεία. Οπότε προσπαθεί να πλουστεύσει την εφαρμογή των προγραμμάτων πλαίσιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτό πρέπει να γίνει αποδεκτό. Πρόθεσή μου είναι να μην περιγράψω λεπτομερώ την προσέγγιση του ελεκτικού συνεδρίου. Όμω, όσον αφορά τα αποτελέσματα των δοκιμών δειγμάτων 97 συναλλαγών στην έρευνα, διαπιστώσαμε ότι 39% αυτών επηρεαζόταν από σφάλματα. Αυτό δεν είναι ικανοποιητικό. Πιθανότερο σφάλμα που υπολογίσαμε όσον να εσωτερικών πολιτικών και έρευνα είναι 1,4%. Τα απορίσματά μας ε, χωρίζονται σε δύο τομείς. Πρώτος, της των πληρωμών βάσει των ελέγχων. Συμπεράναμε ότι οι πληρωμές δεν εμπειρήχαν υλικά σφάλματα. Όμως υπήρχε σημαντικό επίπεδο σφαλμάτων και συχνότητα σφαλμάτων στις ενδιάμεσες τελικέ πληρωμέ του ε, προγράμματο πλαισίου 6 και 7. Και μετά είναι πώ λειτουργούσαν τα εποπτικά ε, συστήματα. Συμπεράναμε ότι τα συστήματα εν μέρη ήταν αποτελεσματικά και μόνο. Παραδείγματο χάρη για, τις, για τους ελέγχους που κάναμε τις αξιώσεις και για τους δικαιούχους για το REACH ε, υπήρχε ανεξάρτητη πιστοποίηση συγκρίναμε τους ελέγχους μας με το πιστοποιητικό που έδωσε ο ανεξάρτητος ελεγκτικός φορέας. 27 περιπτώσεις ο ανεξάρτητος ελεγκτής για το ΡΙΤΣ δεν είχε ε, τεκμηριωμένη άποψη και εντοπίσαμε σφάλματα. Σε 14 περιπτώσεις τα σφάλματα είχαν σημαντικές οικονομικές συνέπειες. Οπότε συστήνουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εντατικοποιήσει τη δράση για να ευαισθητοποιήσει τον εξάρτητου φορεί ελέγχου για του κανόνε για την επιλεξιμότητα των δαπανών. Σημείωσα με τα χαρά στι απαντήσει τη κυρία Κικέν Κουίν ότι προτίθεται πράγματι να δραστηριοποιηθεί στον τομέα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κατά δέντα. Δεύτερη σύστασή μα είναι η εξή. Οι Γενικέ Διευθύνσει Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να μάθουν από τι καλέ πρακτικέ τη Γενική Διευθύνσεω ΙΜΦΣΟ στον ε, τομέα των εκτονιστέρων ελέγχων. Και τέλο, θα ήθελα να εκφράσω τι ευχαριστίε μου προ την κυρία Μέρα Γιώργεν Κουίν, την Επίτροπο και του συναδέλφου τη για την επικοδομητική συνεργασία μα. Διότι αυτό δεν διευκολύνει μόνο το έργο του ελεκτικού συνεδρίου, αλλά εξυπηρετεί τη βελτίωση τη διαχειρήσεω τη χρηματοδοτή των ερευνητικών προγραμμάτων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο τέλο Νοεμβρίου του 2011, το νομοθετικό πακέτο τη του επομένου προγράμματο πλαισίου Horizon 2020 παρουσιάστηκε και υποβλήθηκε. Εμπεριέχει αυτό το πρόγραμμα διάφορε νέε ιδέε όσον αφορά την ερευνητική πολιτική και τη μετοδότηση αυτή και οι συνάδελφοί μου και εγώ ήδη αναλύουμε δεόντω αυτά τα μέτρα για να τοποθετηθούμε όσον αφορά του κανόνε για τη συμμετοχή και διάδοση αυτών των προγραμμάτων όπω προτείνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όπως ήδη έχει ζητηθεί από το Συμβούλιο τις αρχές ε, του έτους. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Συγητή, τα αγαπητοί κυρίες και κύριοι, μέλη της Επιτροπής, θα ήθελα στο τέλος να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πρόσκλησή σας και για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ. Κύριε Μπάρκο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίασή σας στον το έργο του Ελεκτικού Συνεδρίου και θα ήθελα να δώσω το λόγο στην Επίτροπό μας, την κυρία Κέγκεν Κουίν. Απαντήσατε στις ερωτήσεις της Επιτροπής και εκ μέρους όλη τη Επιτροπής θα ήθελα να σα ευχαριστήσω για αυτό και έτσι θα έχουμε αρκετό χρόνο για τα μέλη της Επιτροπής ε, να συμμετάσχουν στη συζήτηση, να θέσουν κάποιες ερωτήσεις. Και γι' αυτό θα ήθελα να σα παρακαλέσω να κάνετε με σύντομη ε, δήλωση, κυρία Επίτροπε. Καλώς ήρθατε στην Επιτροπή. Σας ευχαριστώ πολύ και σας συγχαίρω και για τον ορισμό σας ε, ως Πρόεδρο της Επιτροπής. Αγαπητοί συνάδελφοι, η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση είναι ένα από τα δικά μου καθήκοντα και προτεραιότητα και για να δημιουργηθεί και απασχόληση και θέση εργασία σίγουρα η χρηματοδότηση πρέπει να είναι ελκυστική και να είναι δυνατό να έχουν πρόσβαση σε αυτήν εταιρείε, πανεπιστήμια αλλά και άλλα ερευνητικά ιδρύματα. Σήμερα βρίσκομαι εδώ για να απαντήσω σε κάποιες παρατηρήσεις ιδίως ε, της έκθεσης του 2010 του Ελεκτικού Συνεδρίου και να απαντήσω και στα ερωτήματα των βουλευτών σε σχέση με την έκθεση αυτή. Να σημειώσω με πολύ χαρά ότι δεν υπάρχει ουσιαστικά ε, διαφωνία μεταξύ Επιτροπής και Συνεδρίου. Είναι παρόμοια ανάλυση που κάνουμε και εμείς της κατάστασης ε, και αντίστοιχα και τα αποτελέσματα των δικών μας ελέγχων. Οι δύο συστάσεις του Ελεκτικού Συνεδρίου έγιναν αποδεκτές και θα εφαρμοστούν. Κάτω από το 2% είναι το ασχετικό ποσοστό. Ο συντελεστή αυτή όμω για τι ε, ενδιάμεσε και τελικέ πληρωμέ για τα προγράμματα πλαίσιο είναι υψηλότερε, κάτι αντίστοιχο με τα προηγούμενα χρόνια. Τι μπορούμε να κάνουμε για να μειώσουμε αυτό το ποσοστό σφάλματο. Δύο δυνατότητε. Πρώτον, περαιτέρω διορθωτικά μέτρα ή μέτρα για να αποφύγουμε σφάλματα Είδαμε ποια είναι τα ε, όρια της προστρατηγικής, άρα θέλουμε να κάνουμε πιο απλό το σύστημα, ώστε να μην είναι τόσο εύκολο να γίνουν σφάλματα. Θα ξέρετε ότι το μοντέλο χρηματοδότησης του πρόγραμματος πλαισίου βασίζεται εν γέννη στην επιστροφή ε, του κόστους, του πραγματικού κόστους των συμμετεχόντων. Όπως λέει το συνέδριο, αυτό το μοντέλο χρηματοδότησης ε, δυστυχώς ε, χαρακτηρίζεται από επανειλημμένα σφάλματα. Θα πρέπει λοιπόν ε, να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις. Κάποια μη επιλέξιμα στοιχεία, όπως ο ΦΠΑ, θα πρέπει να αφαιρεθούν. Βέβαια, αυτό δεν το κάνουν πάντοτε οι δικαιούχοι, αλλά με την απόφαση του Ιανουαρίου του 2011 πλουστεύσαμε ακόμη περισσότερο τους κανόνες του 7ου προγράμματος ε, πλαισίου. Πρώτα απ' όλα, οι συμμετέχοντες τώρα μπορούν να υπολογίζουν το κόστος προσωπικού ως ε, μέσο κόστος ε, βάσει του κόστους μισθοδοσίας ε, στους καταστατικούς λογαριασμούς. Επίσης υπάρχει μια καταποκοπή χρηματοδότηση για τους ιδιοκτήτες μικρομεσαίων επιχειρήσεων ή άλλους που δεν λαμβάνουν μισθό. Επίσης το Μάρτιο Έχουμε μια επιτροπή συμψηφισμού ε, που θα βελτιώσει την ασφάλεια δικαίου και θα εξασφαλίσει την ισότιμη μεταχείριση των συμμετεχόντων, ώστε οι θεμητέ προσδοκίε του να γίνονται σεβαστέ όταν έχουν συναλλαγέ με τι υπηρεσίε τη Κομισιόν. Εμεί κάναμε ό,τι μπορούσαμε εντό των ορίων ε, του χρηματοοικονομικού και του χρηματοοικονομικού πλαισίου και ελπίζω όλα αυτά να είναι θετικά και να μειωθεί και το ποσοστό ασφάλματο, τα περιθώρια ασφάλματο. Τώρα θα πρέπει να κεντρωθούμε στο μέλλον. Βασική αρχή μα είναι η απλούστευση και αυτό είναι και στο πλαίσιο του ορίζοντα 2020 και της αναθεώρησης του δημοσιονομικού κανονισμού. Ε, στον ερευνητικό κόσμο οι διάφοροι εμπλεκόμενοι μας είπαν ότι η απλούστευση με το να έχουμε output-based ε, funding ή κατά κοπήν ε, μόνο ποσά, αυτό θα καταστήσει τη χρηματοδότηση λιγότερο ελκυστική γιατί υπάρχει μεγαλύτερο πεθόριο κινδύνου. Θεωρούν λοιπόν ότι απλουστευμένο σύστημα ένα προσταμένο σύστημα θα ήταν πιο ελκυστικό για τη χρηματοδότηση της έρευνας. Ουσιαστικά χρησιμοποιείται η ίδια μέθοδος με αυτή που χρησιμοποιείται στη ΣΥΠΑ και ε, στα κράτη-μέλη. Για να μην έχουμε πολυματικά σφάλματα, ε, θα συνεχίσουμε να ελέγχουμε την κατάσταση. Σε ό,τι αφορά επίσης ανακτήσεις ποσών ή ε, άλλα μέτρα θα συνεχίσουν να ισχύουν και επίσης θα εφαρμόσουμε και την σύσταση του συνεδρίου να έχουμε και εκ των προτέρων ελέγχου, περισσότερο βάσει τη εμπειρία που έχουμε συγκεντρώσει. Αλλά θα πρέπει να υπάρχει και μια θετική σχέση κόστου κόστους-οφέλους για του ελέγχου αυτού και για τους δικαιούχου αλλά και για την Κομισιόν. Ταυτόχρονα όμω θα πρέπει να παραμείνει η ελκυστικότητα τη όλη πολιτική. Ψηφίσατε τον Νοέμβριο του 2010 την έκθεση Καρβάλιο και εκφράσατε ανησυχίε ότι το τρέχον σύστημα και πρακτική τη διαχείριση του 7ου προγράμματο πλαισίου είναι ιδιαίτερα προσανατολισμένη προ τον έλεγχο. Άρα έχουμε μικρότερη συμμετοχή και λιγότερο οικιστικό ερευνητικό πεδίο μεταξύ άλλων. Συμφωνούμε με το Κοινοβούλιο ότι είναι ανάγκη να υπάρξει μεγαλύτερο έλεγχο αλλά και μεγαλύτερη εμπιστοσύνη και σα ευχαριστούμε για την υποστήριξή σα. Οι δικέ μου υπηρεσίε αλλά και εγώ προσωπικά νομίζω ότι έχουμε εξαντλήσει δυναμικό απλούστευση απλούστευσης υπό το νομικό πλαίσιο ε, του τρέχοντος προγράμματος πλαισίου και στο πλαίσιο του δημοσιονομικού κανονισμού. Θέλουμε να υπάρχει σχέση κόστος ωφέλους, αλλά θέλουμε να είναι και ελκυστικό ε, το κλίμα για τις επενδύσεις ε, στην έρευνα και τη χρηματοδότηση της έρευνας. Αφού λοιπόν έχουμε απλουστεύσει, έχουμε όσο, απλουστεύσει όσο μπορούσαμε, θα μπορούσαμε να μειώσουμε το περιθώριο σφάλματος με μεγαλύτερη ανατροφοδότηση για να δούμε ποια είναι τα πιο συχνά σφάλματα και πώς μπορούν αυτά να αποφευθούν. Και αυτό το feedback θα το απευθύνουμε και στους εξωτερικούς ελεγκτές αλλά και στους συμμετέχοντες είναι μια προσέγγιση την οποία το ελεγκτικό συνέδριο αναφέρει στις συστάσεις του και οι υπηρεσίες μου μου ζήτησαν να προχωρήσω προς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα, πώς μπορούμε να τα καταφέρουμε καλύτερα στο πλαίσιο του ορίζοντα 2020 που είναι και πραγματική τομή σε σχέση με το παρελθόν. Διατηρούνται τα καλύτερα τα στοιχεία του πρόγραμματος πλαισίου, αλλά αλλάζουμε και θέλουμε να επιφέρουμε ακόμα μεγαλύτερη απλούστευση Όλοι οι χρηματοδότηση, τα χρηματοδοτικά μέσα τη έρευνα και τη καινοτομία θα μπουν στο ίδιο πλαίσιο, το πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα. Ε, και εκεί θα μπουν και οι δραστηριότητες καινοτομία. Ο Horizon 2020 επικεντρώνει στο να δημιουργήσει καινοτόμα σχέδια και υπηρεσίες ε, μέσα από την έρευνα. Η απλούστευση λοιπόν είναι στο επίκεντρο όλης αυτής της προσπάθειας για να μειώσουμε το άκτος των συμμετεχόντων αλλά και τα σφάλματα που γίνονται με τη χρηματοδότηση έρευνα και της ανάπτυξης. Έχουν γίνει πολλές προσπάθειες για την απλούστευση των κανόνων από την στιγμή που υποβάλλονται οι προτάσεις για σχέδια μέχρι να φτάσουμε στο στάδιο της πληρωμής. Θα σας πω ποια στοιχεία θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερη απλούστευση. Ενία δέσμη μέτρων που θα καλύπτει όλες τις συνιστώσεις του ορίζοντα 2020 σύμφωνα και με τον αναθεωρημένο δημοσιονομικό κανονισμό. μένει κανόνε ό,τι αφορά και τι λογιστικέ πρακτικέ των συμμετεχόντων. Δηλαδή, ε, κόστο μονάδα ε, και. Αυτό είναι το κόστος το οποίο θα χρησιμοποιείτε. Μία, ε, μόνο ένα συντελεστής, αντικατάσταση των τεσσάρων μεθόδων υπολογισμού ε, των πάγιων και έμεσων εξόδων με ένα μόνο καταποκοπή ποσό. Μειώνεται έτσι σημαντικά το περιθώριο σφάλματο, καθώ επίση αναθεωρημένη στρατηγική ελέγχων ε, με επικέντρο την ε, πρόληψη για να ακολουθήσουμε τις, αυτά που μας ζήτησαν από το Κοινοβούλιο σε ό,τι αφορά τον εξωτερικό έλεγχο. Στόχος μας είναι να φτάσουμε στο 2% περιθώριο σφάλματος, αλλά να διατηρήσουμε μια ελκυστική διεθνώς ερευνητική πολιτική. Αυτός ο στόχος θα παραμείνει, αλλά με τις προτάσεις αυτές και με τα στοιχεία της απλούστευσης που περιλαμβάνει ο αναθεωρημένος δημοσιονομικός κανονισμός, νομίζω ότι με όλα αυτά θα σημειώσουμε πολύ μεγάλη πρόοδο για να έχουμε μια απλή δίκαιη χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να έχουμε και την ε, καλύτερη ε, δυνατή σχέση Κόστου ωφέλου. Είναι κάτι το οποίο αξίζουν οι φορολογούμενοι, δηλαδή να έχετε μεγαλύτερη δυνατή απόδοση η επένδυση που κάνουν. Ολοκληρώνοντα, κύριε Πρόεδρε, να σα ε, διαβεβαιώσω για μια ακόμη φορά ότι είμαστε δεσμευμένοι υπέρ τη χρηστή οικονομική διαχείριση, αλλά και υπέρ ε, τη ε, αριστεία στην έρευνα, της πρόσβασης ε, στην ε, έρευνα, ώστε να έχουμε μεγαλύτερη ανάπτυξη και απασχόληση. Είμαι βέβαιη ότι μπορούμε να βρούμε την ισορροπία μεταξύ των στόχων αυτών και ελπίζω και οι στόχοι αυτοί οι δύο να ολοκληρωθούν και όσο διαρκεί το νυν πρόγραμμα πλαίσιο, αλλά και μετά στη συνέχεια με τον ορίζοντα 2020. this Νομίζω ότι μπορούμε πραγματικά να συσχετίσουμε την ε, χρηστή χρησιμοποίηση των χρημάτων και να έχουμε παρόλα αυτά καλά αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο στον εισηγητή, τον Κρίστο Φιάλνα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο <clears throat> και όσους ε, εργάστηκαν πάνω στην προετοιμασία αυτού του κεφαλαίου της ε, έκθεσης, γιατί πρόκειται για ένα βασικό τομέα της ε, κοινοτικής πολιτικής για έρευνα και καινοτομία και είναι ένας τομέας που αφορά το μέλλον. Εγώ θα αναφερθώ σε δύο στοιχεία στην παρέμβασή μου αυτή. Το πρώτο που θα ήθελα να αναφώ είναι τα συμπεράσματα του συνεδρίου όσον αφορά τον, τακτικό, την τεχνική μορφή των πληρωμών και το δεύτερο εκείνο που αφορά τις καινοτομίε. Ε, να σα πω την αλήθεια, ήμουν προετοιμασμένο και για ένα τρίτο θέμα, το θέμα της απλούστευσης. Αλλά είμαι αρκετά ευτυχής με αυτό που άκουσα. Και αντί να απαριθμίσω όλες τις ερωτήσεις στις οποίες δόθηκαν απαντήσει, θα ήθελα εκ στιγμή να σα ευχαριστήσω για τι προσπάθειε που καταβάλατε για το θέμα της απλούστευσης, γιατί αυτό είναι κάτι που όλοι μας θεωρούμε σημαντικό. Τώρα για το πρώτο σημείο. Ε, τακτικός χαρακτήρας των πληρωμών. Το συνέδριο αξιολογεί ότι το περιθώριο ασφάλιμπτος είναι 1,4%. Το 70% όμως των δαπανών για το 7ο πρόγραμμα δράσης εφαρμόζεται ε, βάσει της αρχής της προχρηματοδότησης. Ξέρουμε όλοι ότι η προκατατική αυτή χρηματοδότηση απαιτεί την συμμόρφωση με λίγους μόνο κανόνες εν αντιθέσει προς την χρηματοδότηση κατά τη διάρκεια του προγράμματος ή εκ των υστέρων και γι' αυτό είναι δύσκολο να κάνει κανένα σφάλμα στην προχρηματοδότηση. Γι' αυτό θα ήθελα να ρωτήσω την Επιτροπή να ξέρει ποιο θα ήταν το σφάλμα εάν εκεί γινόταν η χρηματοδότηση εκ των υστέρων κατά τη διάρκεια του, ε, του, του προγράμματος. Δηλαδή, εάν το 70% δεν προχρηματοδοτεί ποιο θα ήταν το ποσοστό σφάλματος στα διάφορα προγράμματα πλαίσιο. Επίσης, με ενδιαφέρει να ακούσω τη σκέψη σας για το ποιο είναι πιο σημαντικό. Ένα ποσοστό σφάλματος με ή χωρίς προχρηματοδότηση. Και βέβαια και γιατί, γιατί και αυτό είναι κάτι που πρέπει να καταλάβουμε. Επίσης, το συνέδριο στην παράγραφα 649 λέει ότι το σύστημα ελέγχου και εποπτείας ήταν μόνο μερικώς αποτελεσματικά και γι' αυτό θέλω να ακούσω εδώ και το ηλεκτρικό συνέδριο και την Επίτροπο να σχολιάσουν και να μας δώσουν τις απόψεις τους όσον αφορά τις πιο σημαντικές ατέλειες των διαδικασιών επιτήρησης. Και τέλος, ποια είναι βέβαια τα συγκεκριμένα μέτρα που παίρνει ή θα πάρει η Κομισιόν για να εξασφαλίσει αποτελεσματικό σύστημα ελέγχου ή εποπτείας. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας. Επίσης θα ήθελα να συζητήσω μαζί σας τα αποτελέσματα που μας δίνει το συνέδριο όσον αφορά το πόσο μπορεί κανένας να βασιστεί στην διαχείριση, γιατί φαίνεται ότι η Κομισιόν βασίζει την αξιολογήσή της στο ότι όλα τα σφάλματα που βλέπουμε θα διορθωθούν. Μετά όμως λέει το συνέδριο ότι η Κομισιόν δεν εξασφαλίζει συστηματικά την ε, διόρθωση όλων των σφαλμάτων. Άρα αυτή η υπόθεση δεν είναι τελικά αληθής. Και θα ήθελα να πω ότι το θέμα είναι αρκετά σημαντικό, γιατί το ποσοστό σφάλμα της, σφάλματος συγγνώμη, της Κομισιόν είναι ένα σημαντικό, για να μην πω το πιο σημαντικό στοιχείο, στο κατά πόσο θα πρέπει να έχουμε επιφύλαξη μέσα στα πλαίσια του έκθεση για την ετήσια ε, δραστηριότητα. Και εάν το, η βάση υπολογισμού δεν είναι σωστή, τότε οι πληροφορίες που παίρνουμε εδώ δεν είναι επίσης σωστές. Και υπάρχει συγκεκριμένα η υπόθεση αυτή στα πλάσια της ε, ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων από την Αρμόδια Γενική Διεύθυνση που θα ήθελα να αναφέρω. Γιατί το συνέδριο λέει ότι το... η επιφύλαξη που υπήρχε για το έκτο πρόγραμμα δράσης έχει αρθεί παρόλο που το ποσοστό σφάλματος ξεπερνάει το κατόφλιο του 2%. Και η Κομισιό απαντά ότι η άρση αυτής της επιφύλαξης έγινε κατόπιν εις βάθους ανάλυσης και βάσει των πιο προσφάτων στοιχείων που επιβεβαιώνουν ότι το ποσοστό σφάλμα θα, θα πρέπει να μειωθεί κάτω του 2% μέχρι τα τέλη του έτους. Δεν ήταν λοιπόν νομίζω εδώ πολύ συνετή η στάση της Κομισιόν. Έχουν την εντύπωση ότι οι υπηρεσίες Κομισιόν ίσως είναι υπερβολικά αισιόδοξε. Λοιπόν κυρία Επιτροπέ, θεωρείτε ότι η έκθεση του Γενικού Γραμματέα στα πλαίσια της ετήσιας έκθεσης είναι σύμφωνη με αυτά που ε, εσείς θέλετε. Λέτε το ποσοστό θα πρέπει να μειωθεί κάτω του 2%. Λοιπόν, αυτό είναι κάπως αντίθετο με αυτό που προσπαθεί να μας πει το συνέδριο και αυτό που μας λέτε εσείς. Θα ήθελα παρακαλώ να μου αναπτύξετε αυτό το σημείο. Και να έχετε επίσης κατά νου ότι η επιφυλάξη του συνεδρίου όσον αφορά την συνθετική έκθεση της ε, Κομισιόν στην συνθετική αυτή έκθεση η Κομισιόν ενημερώνει το Κοινοβούλιο και ποια είναι η σχέση της έκθεσης αυτής με την έκθεση του Γενικού Γραμματέα. Αυτές είναι οι ερωτήσει μου προς το Ελεκτρικό Συνέδριο και προς την Κομισιόν. Ελπίζω να μην είναι πολύ δύσκολες. Και... Ε, Ευχαριστώ κύριε Σιγητά. Η Επίτροπος ε, κυρία Γεώργια να θέλει να απαντήσει αμέσως, μπορεί να πάρει το λόγο. Ε, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ξεκινήσω με τα ποσοστά σφαλμάτων. Καταρχάς, για το πρόγραμμα πλαίσιο 6 το ποσοστό που εντοπίστηκε ετήσια είναι περίπου 3,5% και μειώθηκε στο 2,4% περίπου μετά από ανακτήσεις και διορθώσεις. Σε πολιτή βάση ήταν αυτά λαμβάνονται υπόψη. Για το πρόγραμμα πλαίσιο 7 το ποσοστό σφάλματο δεν έχει καθοριστεί επί κανονικού δείγματος. Επί περιορισμένου σχετικά δείγματο που επικεντρώνεται επί νέων ή μη ελεγχθέντων δικαιούχων αναμένεται χαμηλότερο επίπεδο σφάλματο, Λίγο πάνω από το 4% ετησίω. Δεν είχαμε αρκετό χρόνο ακόμα να δούμε ποιες είναι οι πλήρες συνέπειες των διορθώσεων και των ανακτήσεων σε πολιετή βάση, ούτε και πιο σημαντικό αυτό τα αποτελέσματα των μέτρων απλούστευσης που προανέφερα. Τώρα το ποσοστό σφάλματος θα ήταν υψηλότερο αν δεν λαμβάναμε υπόψη την χρηματοδότηση στη δειγματοληψία. Το δείγμα ελέγχου που χρησιμοποιείται από το ελεγκτικό συνέδριο για να τοποθετηθεί όσον αφορά την έρευνα και την εσωτερική πολιτική συμπεριλαμβάνει προχρηματοδότηση, ε, ενδιάμεσες πληρωμές και τελικές πληρωμές. Όμως έλεγχοι που διεξάγονται την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο δικό της αντιπροσωπευτικό δείγμα που καλύπτει μόνο προσωρινές τελικές πληρωμές δείχνει ότι ο ποσοστό σφάλματος είναι παρόμοιο με αυτό που βρίσκει το ελεκτικό συνέδριο. Τι προβλέπουμε για το 2011 και 2012 όταν είναι ακόμα μεγαλύτερα τα προγράμματα εργασιών δεν αναμένονται δραματικές αλλαγές και είμαι αισιόδοξη. Πιστεύω ότι θα δούμε μείωση του ποσοστού σφάλματος λόγω των μέτρων απλουστεύσεως που εισήχθησαν το 2011. Επιπλέον, το 2012 θα ενισχύσουμε προσπάθειες για προσανατολισμό παροχή συμβουλών στους συμμετέχοντες και τους ελεγκτικούς φορείς για να αποφύγουμε τα σφάλματα. Να κάνουμε και αυτό που είπε ο Σμπάλκο, να αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση όσον αφορά τα συχνότερα σφάλματα και να ασφαλίσουμε καλύτερη κατανόηση των διαφόρων κανόνων που διέπουν αυτές τις εργασίες. Δεν ξέρω αν θέλετε να απαντήσω το δεύτερο ερώτημα ή να απαντήσει ο κύριος Μπάλκο τώρα, κύριε Πρόεδρε. Α, καλώς. Όσον αφορά την εξοπιστία των πιστοποιητικών ελέγχου. Όσον αφορά τα πιστοποιητικά ελέγχου, ήδη έχουμε λάβει τα μέτρα για βελτίωση της αποτελεσματικότητας αυτών όπως τα πορίσματα των ε, ελέγχων να τροφοδοτούνται στους δικαιούχους, να δημοσιεύουμε πληροφορίες και οδηγίες και δημιουργώντα υπηρεσία για έρευνες ε, ε, ούτω ώστε να δίδονται απαντήσεις του ελεγκτικού φορεί. Τα προβλήματα που εντοπίσαμε αφορούν κυρίω το πρόγραμμα πλαίσιο 6 και τα πιστοποιητικά ελέγχου. Για το πρόγραμμα πλαίσιο 7, ο αριθμό των πιστοποιητικών που ζητήθηκε μειώθηκε δραστικά όσον αποτέλεσμα των μέτρων πλούστευση και η μεθοδολογία άλλαξε για την βελτίωση των αποτελεσμάτων. Πρόοδο προφανώ θα παρακολουθείτε εκ του σύνεγγυ φέτος, το 2012, βάσει των αποκτηθισών εμπειριών για την εφαρμογή του προγραμμάτου πλαισίου 7 θα ενισχύσουμε τις προσπάθειες για να δίνουμε οδηγίες στους συμμετέχοντες και στους διάφορους ελεγκτές που χορηγούν τα πιστοποιητικά για την αποφυγή σφαλμάτων σε αφορά τη διαχείριση. Για να υποστηρίξουμε σωστά τα πιστο... τις ε, αξιοπιστίας των διαφόρων ε, διευθυντικών φορέων οι υπηρεσίε μα έχουν ένα κοινό τύπο για τον υπολογισμό των αντιπροσωπευτικών σφαλμάτων και των υπολοιπωμένων σφαλμάτων, των υπολείπων σφαλμάτων, ανανεώθηκε η μεθοδολογία και οι διαφορές που υπάρχουν στη μεθοδολογία θα μειωθούν. Και θέλουμε αρμονισμένη προσέγγιση για την ανάλυση και την κοινοποίηση των πορισμάτων των, των ερευνών που γίνονται όσον αφορά το πρόγραμμα πλαίσιο 7. Ευχαριστώ κυρία Επίτροπε, λέει ο Πρόεδρος. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Μπάλκο του ηλεκτρικού Συνεδρίου, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, ε, κύριε Πρόεδρε. Για να εξοικονομήσω χρόνο για την Επιτροπή σας, θα προσπαθήσω να απαντήσω στον εισηγητή στο ερώτημά του που αφορά τα συστήματα για την αποφυγή και διόθου σφαλμάτων αναφέραμε ότι υπάρχουν δύο δυναμίες. Πρώτη, εκ των προτέρων έλεγχη. Δεύτερη, η πιστοποίηση των ελέγχων. Πρώτον, η εκ των προτέρων έλεγχη. Είναι περιορισμένη η πολιτική επιλογή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όσον αφορά την πιστοποίηση ελέγχων για τις αξιώσεις δαπανών, το ανέφερα αυτό όταν μίλησα προηγουμένως. 33 αξιώσεις ελέγχθηκαν και κάθε πιστοποιητικό που χορηγήθηκε από τον εξάρτητο ελεγκτικό φορέα συμπεριλάβαμε τις παρατηρήσεις μας στη δεύτερη σύστασή μας. Στο σημείο 6.51 Εκεί στη δεύτερη σύσταση αναφέρουμε ότι για να βελτιώσουμε περαιτέρω την αξιοπιστία των πιστοποιητικών ελέγχου εντατικοποιούμε την ε, δράση για να βιστοποιήσουμε τους ελευνητικούς φορείς για την επιξημότητα ε, και τους ενημερώνουμε επίσης και το που δεν έχουν εντοπιστεί οι δαπάνες οι οποίες δεν είναι επιλέξιμες. Και δέχτηκε τις συστάσεις μας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις δύο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπάλκο. Οι συνάδελφοι έχουν το λόγο τώρα. Πρώτη η συνάδελφος Ιβάνοβα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Επίτροπε, επιτρέψτε μου να σας συγχαρώ για την ομιλία σας. Εδώ είμαι, εδώ είμαι. Here. Hello. Uh, I, I must say that... Είμαι πολύ ικανοποιημένη. Όπως και ο συνάδελφος Χέλλον, άκουσα τη λέξη απλούστευση να επαναλαμβάνεται. Αφορούσε ένα από τα ερωτήματά μου αυτό. Αλλά τώρα μου έμεινε ένα σύντομο σχόλιο. Μου άρεσαν αυτά που είπατε. Ελπίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξασφαλίσει ότι θα εφαρμόζονται αποτελεσματικοί έλεγχοι για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της κοινότητας. Δύο ερωτήσεις έχω. Πρώτη, όσον αφορά το πρόγραμμα πλαίσιο Horizon 2020 για έρευνα και καινοτομία, υποστήριξη επιχειρήσεων. Ερώτηση. Περισσότερες λεπτομέρειες μας δίδεται. Ποια ήταν η επιρροή, πώς επηρέασε τις επιχειρήσεις το 2010, διότι είναι βασικό αυτό για μας, ε, για την αναζωγόνηση της ευρωπαϊκής οικονομίας. Η άλλη ερώτηση. Για το μέσο για το διαμοιρασμό του κινδύνου. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική ε, Τράπεζα Επενδύσεων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρησιμοποιούν αυτό το μέσο για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων έρευνα και ανάπτυξη στα πλαίσια του προγράμματο πλαισίου 7 ένα δισεκατομμύριο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ένα δισεκατομμύριο την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Διάβασα εν μέρη την ενδιάμεση αξιολόγηση του μέσου αυτού για το 2010. Εκεί εμπεριείχε το μια σύσταση. Η σύσταση έλεγε ότι η συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σαν ένα πρώτο εργαλείο, διότι υπάρχει αυξανόμενη ζήτηση για αυτή τη χρηματοδότηση. Και αυξανόμενο κίνδυνο υπάρχει όμω για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ταυτόχρονα. Μπορεί να αναλάβει τον κίνδυνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι έτοιμη να αναλάβει αυξημένο κίνδυνο ή όχι. Ποια είναι η άποψή σα για την επιλεξιμότητα, για τα σφάλματα επιλεξιμότητα αυτό συνδέεται με την απλούστευση. Αν υπάρχει σύστημα ε, διάδοσης καλών πρακτικών και αυτό θα συνέβαλε στη μείωση αυτού του είδους ε, σφαλμάτων, ε, κινδύνου σφαλμάτων. Ευχαριστώ κύριε Ιφανό. Θα έλεγα να συλλέξουμε μερικέ ερωτήσεις. Η σωσταστική ομάδα δεν θέλει να βάλει καμία ερώτηση. Ο συνάδελφος Κατζημαρκάκης όμως. Ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επίτροπο για τις απαντήσεις που έδωσε στις ερωτήσεις μας και για την παρουσία της. Θα ήθελα καταρχήν να πω ότι είναι πάρα πολύ καλό από τις αρχές του 2012 η Κομισιόν έχει ενιαία συστήματα ελέγχου των λογαριασμών. Είναι κάτι που είχε ζητήσει πολλές φορές το Κοινοβούλιο. Υπάρχουν διάφορες γενικές διαθέσεις που άσκουν ερευνητική πολιτική, διάφορες υπηρεσίες, και είναι πολύ πιο απλό να έχουμε ένα ενιαίο σύστημα ελέγχου. Είναι και πιο γλίγορος ο έλεγχος αυτός σήμερα. Ε, περνάνε μόνο 380, 338 μέρες ε, μεταξύ της υποβολής της αίτησης και της πληρωμής. Ε, έγκαιρα πληρώθηκαν τα χρήματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ήθελα όμως να κάνω κάποια παρατήρηση. Ε, γιατί σε μια ερώτησή μας δεν πήραμε πολύ συγκεκριμένη απάντηση. Αναφερθήκατε και εσείς στο σύστημα των πόντων, αν θέλετε. Σας το υποβάλαμε αυτό προς έλεγχο. Μας είπατε ότι δεν θέλετε να εισαγάγετε ένα τέτοιο σύστημα, αλλά ε, σε σχέση και με τον ορίζοντα 2020 να δίνετε ε, βραβεία. Η ίδια κατεύθυνση είναι. Αλλά δεν μας λέτε ακριβώς τι θέλετε στις λεπτομέρειες. Και θα ήθελα να ξέρω σε ποιους τομείς και ποιο ποσοστό της χρηματοδότησής σας θα ε, είναι εκείνο το που θα καλύπτεται από τα βραβεία αυτά. Γιατί και με καταποκοπήν ποσά μπορούν πάλι να υπάρχουν απλουστεύσεις. Εσείς είπατε θέλετε να σαγάγετε κάποιες ε, Τέτοιε καταποκοπήν πληρωμέ, αλλά είναι ασαφή η απάντησή σας, δηλαδή ποιο ποσοστό, ποιοι τομεί θα είναι εκείνοι που θα αφορούνται από αυτό. Εγώ θα ήθελα, μια που είσαστε η πρώτη επίτροπος που ήρθατε εδώ, να διαμαρτυρηθώ γιατί δεν έχουμε ακόμα την έκθεση αξιολόγησης μετά από τα τέλη του 2011 τα οποία μας είχε υποσχεθεί η Κομισιόν αυτό το έγγραφο. Είσαστε πρώτες εσείς εδώ και γι' αυτό σε εσά θα διαμαρτυρηθώ. Τώρα μας λένε θα έρθει τέλη του ε, Ιανουαρίου. Αυτό είναι πολύ άσχημο γιατί δεν μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε για την απαλλαγή. αναφέρουμε στην έκθεση αξιολόγηση. Ξέρω ότι δεν φταίτε εσεί, αλλά παρακαλώ να το μεταβιβάσετε αυτό που σα λέω, γιατί πρέπει να έχουμε κάθε ευκαιρία να εξετάζουμε την αποτελεσματικότητα και τη πολιτική έρευνα που πρέπει εσείς λόγω των υποχρεώσεων της συνθήκη της Λισαβόνας να ξέρετε ότι θα την ελέγξουμε και δεν μπορούμε να την ελέγξουμε σωστά. Παρακαλώ λοιπόν να προωθήσετε την πρόταση αυτή στον κύριο Σένατα και στον πρόεδρο Μπαρόζο ιδιαίτερα γιατί δεν έχουν εκπληρώσει μια υποχρέωση που ανέλαβαν. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ κύριε Χαζημαρκάκη. Η συνάδελφος Γκρέσλα έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, πολλά προβλήματα νομίζω μπορούμε να λύσουμε με τον οργανισμό Ορίζον 2020 και ε, εγώ είμαι η συγκήτρια για τον δημοσιονομικό οργανισμό και προσπαθώ κάποια να, πράγματα να καταφέρω. Δεν είναι όμως πολύ απλό αυτό. Ιδίως μα που βλέπω ότι για το θέμα αυτό ο καθένας έχει το δικό του αγαπημένο θέμα και ακολουθεί το δικό του θέμα αυτό μέχρι που να μην υπάρχει τίποτα κοινό με πια. Θα θέλω λοιπόν να μπορώ να πω στου συναδέλφου ότι όλα πάνε πολύ καλά. Θέλω να υποβάλω ένα ερώτημα όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογία. Ακούω φρικτά πράγματα για το Ινστιτούτο αυτό. Εσεί, από δική σα σκοπιά πώ βλέπετε τα πράγματα. Μήπως θα μπορούμε να είχαμε κάποια έτσι ενθαρρυντική έκθεση για την κατάσταση αυτού του Ινστιτούτου. θα ήθελα να ξέρω και πώς είναι εκεί κατανομημένες οι αρμοδιότητες γενικά και μέσα στην Κομισιόν. Ένα αυτό. Δεύτερον, έχουμε να εξετάσουμε σήμερα και μια ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου για τον μηχανισμό εγγυήσεων υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Πολύ επιτυχές το πρόγραμμα αυτό. Πρόκειται για δημοσιονομικά μέτρα, αλλά εσείς ε, ε, έχετε κάποια μέσα για να δώσετε και άλλες εγγύησεις ε, εκτός των ΜΜΕ, εσείς πώς εκτιμάτε την επιτυχία αυτών των μέσων και πότε θα πάρουμε και μια γραπτή έκθεση για να ξέρουμε ότι πραγματικά τα πράγματα πήγαν έτσι όπως έπρεπε να πάνε. Γιατί βέβαια είναι πάρα πολύ δύσκολο να προσπαθώ να ε, καταλήξω σε κανόνες χωρίς να ξέρω ποια είναι τα αποτελέσματα μέχρι στιγμής. Ευχαριστώ, πρόεδρος. Ευχαριστώ, κύριε Γκρέσερ. Ο Παύλου Ρουμπίχ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Αναφέρθηκε ήδη το γεγονός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες ακριβώς ε, λόγω της κρίσης έχουν προβλήματα, γιατί δεν έχουν και την απαραίτητα ρευστότητα πάντα. Ρωτάω λοιπόν, τι γίνεται με τα προγράμματα Eurostars και ΕΡΕΚΑ. η εξέλιξη εκεί για περισσότερη ευστότητα υπέρ των ερευνητικών δραστηριοτήτων έχει προχωρήσει. Πρώτα σε ευχαριστώ κύριε Ρουμπίχ. Πρωτού σα ε, δώσω το λόγο κύριε Επίτροπε για να απαντήσετε στι ερωτήσει αυτέ. Έχω κι εγώ μια ερώτηση. Αναφερθήκατε στο θέμα του φόρου προστιθέμενης αξίας, με... απάντηση δηλαδή στην ερώτηση 16 είναι πολύ καλό για αυτούς που ζητάνε επιδοτήσεις ότι τώρα θέλετε να συμπεριλάβετε τον ΦΠΑ στο επιλέξιμο κόστος. Μπορείτε να μας πείτε πώς εκτιμάτε το θέμα των διαφορετικών ΦΠΑ στα κρατη κατά πόσον εκεί υπάρχουν κάποιες επιπτώσεις ανακατανομής ή εξεδοτηρώνονται αυτές. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Επίτροπος έχει το λόγο. Παρακαλώ. Thank you, uh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, το έθεσε και ο Αντιπρόεδρος ε, και εσείς και η κυρία Γκρέσλε και κάποιοι άλλοι. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι όπως γνωρίζουμε όλοι η σπονδυλική στήλη της ευρωπαϊκής οικονομίας και είναι ένα θέμα που απασχολεί πολύ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρέπει να πω όμως και την Κομισιόν. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορούν να συμμετέχουν οι, Ευρω... οι ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις και συμμετέχουν ε, σε αυτό το πρόγραμμα στήριξη της έρευνας. Νομίζω ότι αν το δείτε αντικειμενικά θα δείτε ότι έχουμε πράγματι σημειώσει πρόοδο και έχουμε αναβαθμίσει τις προσπάθειές μας για να φτάσουμε στο 15% που στους θεματικούς τομείς έχουμε εγγυηθεί. Επίσης, ε, ξεκινήσαμε πολύ πρόσφατα μια νέα πρωτοβουλία ε, σε ό,τι αφορά και το δημοσιονομικό μέσο επιμερισμού των κινδύνων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα δώσει 120 εκατομμύρια συμμετοχή με και αναμένεται να έχουμε ένα δις περίπου δάνεια για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ο Ορίζον 2020 βάζει στο επίκεντρο της στήριξης μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μαζί με τις προσδοκίες για το 15% έχουμε και τις εταιρικέ προκλήσεις και τις διάφορες τεχνολογίες που μπορούν να διευκολύνουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά θα έχουμε και ένα νέο μέσο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που βασίζεται σε ένα μέσο το οποίο είχε εισαχθεί ε, στις ΕΠΑ, το SPIR. Πολλά, μέσα, πολλά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής σας και άλλοι από την Επιτροπή Τρέμου το έχουν αναφέρει, αυτό το αμερικανικό αντίστοιχο ε, μέτρο. Θα έχουμε και με την υποστήριξη μέσω επιχειρηματικού κινδύνου και για τις νεοσυσταθείς εταιρείε και για τις μεροκαμιστές επιχειρήσεις στήριξη αλλά θα έχουμε ωφέλεια και από αυτά τα πολύ ριζικά μέτρα πλούστευση που εισάγουμε το 2000 ε, και τον οριζόντα 2020. Παναλαμβάνω και σα ε, διαβεβαιώνω ότι εξίσου, σημαντικό, ε, εξίσου σημαντικές είναι οι μικρομεσαίε επιχειρήσεις όχι μόνο για το κοινό και για την Κομισιόν. Τώρα, να απαντήσω σε αυτό που είπε η κυρία Γκρέσλε για την αξιολόγηση των χρηματοοικονομικών εργαλείων. Το καλύτερο παράδειγμα που έχουμε είναι η ανεξάρτητη έρευνα για το RSS, RSF ήταν πάρα πολύ θετικό το πόρισμα και καλό είναι να υπάρχουν εξάρτητες αξιολογήσεις γιατί έτσι έχουμε και μια αντικειμενική εικόνα. Μετά λοιπόν το αίτημα και του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και με βάση όσα μας έδειξε η ενδιάμεση αξιολόγηση του RSFF έχουμε την συμφωνία που υπογράψαμε στις 15 Δεκεμβρίου και θα έχουμε ένα νέο ειδικό μέσο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις Risk Sharing Instrument, RSI, σας το είπα και πριν. Έχουμε λοιπόν αυτό το νέο μέσο, το οποίο θα εφαρμοστεί με εταιρική σχέση επιμερισμού κινδύνων μαζί με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων. Αναμένεται λοιπόν να έχουμε μόχλευση 8 φορές ε, της συμβολής ε, της Ένωσης, 120 εκατομμύρια, σας είπα το ποσό και πριν. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να πούμε ότι η Κομισιόν θεωρεί ότι η επιχειρησιακή και χρηματοοικονομική αναφορά που ζητήθηκε αλλά και δίνεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων πάρα πολύ σημαντική. Μα δίνει στοιχεία ώστε να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε και την παρακολούθηση και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση. Απαντώ πάλι στην κυρία Γκρέσλι. Νομίζω λοιπόν ότι το RSFF, όταν ήμουν στο Κοινοβούλιο αλλά και εκτός Κοινοβουλίου, ε, πάντα λέω ότι ήταν μια πολύ μεγάλη επιτυχία, πολύ μεγαλύτερη από αυτό που μπορούσε κανείς να φανταστεί όταν ε, πρώτο έγινε η συμφωνία μεταξύ Κομισιών και Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων. Σε ό,τι αφορά αυτό που είπε ο κ. Χατζημαρκάκης, για αυτούς τους πόντους, τα μπόνους. Δεν μπορούμε βέβαια να πούμε αυτή τη στιγμή στην ε, ΧΥΠΣΥΠΕ το τομέα θα έχουμε αυτή τη τα κτλ. Αλλά ε, αυτό τη ε, η βάση που είχαμε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχουν κάποιε εταιρικέ προκλήσει. Καλούμε την ερευνητική κοινότητα λοιπόν να ανταποκριθεί στην πρόκληση, στι προκλήσει και βάζουν και μια τιμή. Αυτό κάναμε και ήταν πολύ επιτυχημένο στην Ευρώπη αλλά και σε άλλες χώρες στον κόσμο. Δεν έχουμε λάβει όμως αποφάσεις γιατί ορίζοντα το 2020 ναι. δημοσιεύθηκε μόλις πριν τα Χριστούγεννα. Έκανα μια αρχική παρουσίαση και στο Συμβούλιο Υπουργών και στο Κοινοβούλιο. Μπορούμε όμως νομίζω τώρα να το συζητήσουμε όσο προχωρεί αυτή η διαδικασία και στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο. Ίσως υπάρχουν απόψεις για το πώς μπορεί να γίνει, ποιου τόμεις πρέπει να στοχεύσουμε. Νομίζω θα είναι πολύ χρήσιμη η συζήτηση, πολύ επικοδομητική και ελπίζω να είναι και ιδιαίτερα ζωντανή σε ό,τι αφορά τον τομέα αυτό για να απαντήσω στην κυρία Γκρέσλε σε ό,τι αφορά το EIT. Ε Ήταν πάρα πολύ χρήσιμο, πρώτα απ' όλα η έκθεσή της και όλα τα στοιχεία τα οποία έχουμε λάβει τα λαμβάνουμε πάρα πολύ Είναι ένα θέμα όμως που δεν αφορά άμεσα το δικό μου χαρτοφυλάκι, αλλά την κυρία Βασιλείου. Useful point to be raised with Commissioner Vassiliou, but I will certainly bring the points in relation to what... Θα αναφέρω όμως τα σχετικά στην κυρία Βασιλείου και μάλιστα αυτή την εβδομάδα. Ε, Για το ΦΠΑ είναι το θέμα αυτό. Äh, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για το ΦΠΑ μπορείτε να πείτε κάτι άλλο. Ε, συγγνώμη, Πρόεδρε. Έδωσα ένα παράδειγμα για το ΦΠΑ που είναι ένας τομέας που δημιουργεί, δημιούργησε δυσκολίες κατά το παρελθόν ε, στα μη, στις μη επιλέξιμες δαπάνες σε αυτό το τομέα και για μας η συμπερίληψη του ΦΠΑ στο υπολογίσιμο κόστος θα βοηθούσε να μειώσουμε τα σφάλματα του παρελθόντος που διαπιστώσαμε κατά το παρελθόν και έτσι θα μπορέσουμε να παρουσιάσουμε καλύτερο υπολογισμό στο τέλος και καλύτερη απόκριση. Είναι καλός τομέας αυτός, στον οποίο θα πρέπει να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας και σίγουρα μπορούμε να κάνουμε αυτό που είπε σήμερα ο εισηγητής και αρκετά μέλη τα ανέφεραν άλλωστε. Δηλαδή να έρθουμε σε επαφή με τους ελεκτικούς φορείς που ε, έρχονται σε επαφή με τις εταιρείε και ελέγχουν τις δαπάνες τους. Ε, νομίζουμε ότι αυτό είναι ένα πολύ χρήσιμο τρόπο. Έτσι μπορούμε λεπτομερώς να εξηγήσουμε σε αυτούς τι ακριβώς απαιτείται και πώς ε, μπορούν να βελτιωθούν και πώς μπορούμε να συμμορφωθούμε αυτό που θέλει το ελεκτικό συνέδριο. Δηλαδή να αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση των διαφόρων κύκλων, πώς ακριβώς πρέπει να ανταποκρίνονται. Πώς οι εμπλεκόμενοι λοιπόν πρέπει να κινηθούν για να αποφευθούν τα σφάλματα σφάλματα που λαμβάνουν χώρα στην προετοιμασία των απαντήσεών τους. Όλα αυτά μαζί με τα ριζικά μέτρα απλούστευσης μπορούν να βελτιώσουν την όλη προσέγγιση και προφανώς πρέπει να ακούσουμε προσεκτικότατα αυτά που λέγει και αυτή η Επιτροπή και το Ελεκτικό Συνέδριο. Θα πρέπει να τα λάβουμε αυτά που λέγονται υπόψη και να τα αποκριθούμε θετικά. Και αυτό κάναμε και αυτό προτιθέμεθα να συνεχίσουμε και στο μέλλον. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχει κανένα άλλο από την Επιτροπή μα ζητήσει το λόγο. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στον εισηγητή, εάν το επιθυμεί. Όχι, όχι πρόεδρε. Απλώ θα ήθελα επί τη ευκαιρία να ευχαριστήσω τον Επίτροπο για τι απαντήσει τη. Ιδίω όσον αφορά τα ποσοστά σφάναματο για τα διάφορα προγράμματα πλαίσιο. Ήταν πάρα πολύ σημαντικά αυτά. Και θα ήμουν πολύ ευτυχή βέβαια να μα τα έδινε και γραπτό αν ήταν δυνατόν. για να δούμε τα ε, ποσοστά σφάλματος και για το τελικό και για τα προσωρινά ε, προγράμματα. Σας ευχαριστώ πάντως πάρα πολύ κύριε Επίτροπε, δεν έχω τίποτα άλλο αυτή τη στιγμή. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ κύριε εξ Εξοδόματος του συνόλου της Επιτροπής μας και θα χαιρόμαστε πραγματικά να πάρουμε γραπτές αυτές τις ε, απαντήσεις για τις οποίες ζήτησε ο συγητή μας. Σας ευχαριστώ που ήρθατε εδώ. Ευχαριστώ και το ηλεκτρικό συνέδριο και μπορώ τώρα να προχωρήσω στο επόμενο σημείο της ημερής διάταξης. Ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ηλεκτρικού Συνεδρίου και εδώ υπεύθυνο είναι ο Λαντισλαβ Μπάλκο και η συγκήτρια Ίγκεβορ Κρέσλε. Okay. Jetzt ist äh, eine kurze Unruhe. Wir danken nochmal ganz herzlich, Frau Kommissarin. Θα ήθελα για μια φορά να ευχαριστήσουμε την ε, Επίτροπο Γιώργιαν Κουίν και όπως σας είπα, περνάμε στο επόμενο σημείο. Ο κύριος Μπάλκο για το ηλεκτρικό συνέδριο έχει το λόγο. Ε, thank you very much, Mr. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Dear Madam Reporter, Dr. Gressle, ladies and gentlemen. Ευχαριστώ κυρία Συγγετρία κύριε Πρόεδρε, τιμή για μένα, για μία ακόμη φορά, να παρίσταμε εδώ για δεύτερη φορά και να μιλώ για δεύτερη φορά σήμερα εκπροσωπώντα το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο και να παρουσιάσω την ειδική έκθεση 4 του 2011 όσον αφορά τον έλεγχο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ε, με την δυνατότητα παροχής εγγύσεων όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενο σημείο όλοι γνωρίζουμε τη σημασία που έχει αυτός ο μηχανισμός και για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει που είναι η ραχοκοκαλιά ε, της οικονομίας ευρωπαϊκής ε, που παρέχουν οι μικρομεσαίε επιχειρήσεις 75 εκατομμύρια απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμω πολύ συχνά οι χρηματοπιστωτικέ αγορές και το ξέρω πολύ καλά διότι είμαι πρώην τραπεζίτης οι χρηματοπιστωτικέ αγορέ, έλεγα λοιπόν ενδιαφέρονται πολύ για τις νέε νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις κυρίως αν είναι, κινούνται σε καινοτόμες αγορές. Αντιμετωπίζουν καμιά φορά δυσκολίες για πρόσβαση στην σωστή σε σωστά οικονομικού πόρου και αυτό είναι εμπόδιο για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει είτε να δημιουργηθούν ή να αναπτυχθούν. Άρα ε, πρέπει να υποστηριχθεί ο, ο τομέα των μικρομεσαίων όχι απλώς θεσπίζοντας το κατάλληλο νομικό πλαίσιο, αλλά θα πρέπει να παρέχεται και αναγκαία χρηματοδότηση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ένα από τα εργαλεία για την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και για την πρόσβασή της χρηματοδότηση είναι το μηχανισμό SMAC. Είναι ένα οικονομικό μέσο στα πλαίσια ε, του προγράμματος πλαισίου ΣΥΠ για την οικονομική ανάπτυξη ε, που το διαχειρίζει το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο εκ μέρους της Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής που δίνει εγγυήσεις όσον αφορά τους μεσάζοντες για να για τη δανειοδότηση που παρέχεται από χρηματοπιστωτικού φορεί προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στην ειδική έκθεση παριθμών 4 του 2011 παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα του ελέγχου επιδόσεων όσον αφορά το εργαλείο ΣΜΑΚ, όσον αφορά την αποτελεσματικότητά του και πώς σχεδιάζεται η λειτουργία του και εφαρμογή του και πώς ε, επιτυχάνονται οι στόχοι του. Για δώσω μια ολόκληρη εικόνα και για να σας δώσω γενική εικόνα θα ήθελα να αναφέρω εδώ ότι το μέσο ΣΜΑΚ δεν είναι το μόνο οικονομικό μέσο για... που ελέγξαμε ε, για τις μικροσές επιχειρήσεις Ελέγχουμε τώρα και το μέσο για την οικονομική μηχανική, financial engineering, για μικρομεσαίες επιχειρήσεις που σχηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό ε, Ταμείο ε, Ανάπτυξης και ελέγχεται από άλλο φορέα του, από άλλο συνάδελφο του Ελληνικού Συνεδρίου. Τα βασικά πορίσματα του ελέγχου όσον αφορά το μέσο ΣΜΑΚ συνοψίζονται στο έγγραφο εργασία που συνέταξε η Dr. Grace η γήτρια, όμως δράτω με τις να σας δώσω μια σύντομη επισκόπηση των πορισμάτων του ελεκτικού συνεδρίου και των συστάσεων αυτού. Ε, χρειάζεται σωστό πλαίσιο για τη, ε, για τη λειτουργία αυτού του μέσου. Βελτιώθηκε η δομή δίνοντας κίνητα βασίλου τις επιδόσεις. Όμως καθυστερήσεις σχεδιασμού του μέσου επηρέασαν την χρηματοδότηση κατά το πρώτο έτος και οδηγήθηκε και σε διακοπές όσον αφορά την υποστήριξη σε κάποιους ενδιάμεσους χρηματοδότες. Ε, λοιπόν, δεν είχαμε κάποια πρότυμα για τη δαθμολόγηση σωστής επιλογής των μεσαζόντων. Υπήρξαν δείκτες επιδόσεων. Δεν ήταν ισορροπημένοι αυτοί όμως. Ήταν δείκτες μόνο για εκροές. Τα στοιχεία για τους δείκτες αντιχτύπου, ε, τα στοιχεία για τον διαμόρφωση αυτού του δείκτου είναι δύσκολο να συλλεχθούν που αφορούν την δημιουργία απασχόληση. Και υπάρχει και πρόβλημα συγκρισιμότητα μεταξύ χωρών. γενικά με τις απαιτήσει που προβάλλονται τα αποτελέσματα είναι ικανοποιητικά. Το μέσο ΣΜΑΚ φαίνεται ότι λειτουργεί σχετικά σωστά. Θέλουμε να φτάσουμε 350.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο τέλος του προγράμματος και θεωρούμε ότι είναι εφικτός ο στόχος. Το δάνειο χορηγείται στα πλαίσια του ΣΜΑΚ Τα μισά, τα, μισά, τα μισά δάνεια δίνονται χωρίς εγγύσεις και 12% μόνο από αυτά τα χρήματα θα δίδονται σε ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θέλουν να κινηθούν στις καινοτομίες υπάρχει ε, ένα στοιχείο απόβαρου αν θέλετε. Δίνονται κάποια δάνεια στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δεν ε, πληρούσαν τις όρους για τις εγγυήσεις ή που δεν οδήγησαν στις επενδύσεις. Χρειάζεται να αποδεικνύεται πού πηγαίνουν τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι που δεν γίνεται ξεκάθαρα και χρειάζεται να ελεγχθούν και συμφωνίες με τους μεσάζοντες του σωματοξωτικούς. Γίνονται και συστάσεις για την καλύτερη λειτουργία και επίδοση του μέσου αυτού. Και σε παρόμοια προγράμματα υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο μέλλον. Απευθύνουμε συστάσεις κυρίως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αφορούν όμως και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και το Συμβούλιο υπό την ιδιότητά του που είναι και αυτό νομοθέτης. Συστήνω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ταξής. Στόχος η στόχοι στο νέο πολιτές πρόγραμμα δεν είναι πολύ σαφέστερη από ό,τι στο πρώτερο. όπως ήταν και το 2001 με το 2006, συστήνουμε μελλοντικά προγράμματα να εδράζονται επί σαφούς πολιτικής παρέμβασης, εξετάζοντας την εισρωή και τα αναμενόμενα αποτελέσματα του φάτσε κρόες. Δεύτερον, υπάρχει γενικό πλαίσιο για τη διαχείριση του μέσου ΣΜΑΚ. Όμως, εντοπίσαμε καθυστερήσεις στο σχεδιασμό της προχρηματοδότησης το πρώτο έτος. Συστήνουμε λοιπόν να τελειοποιηθεί η νομική βάση και η συμφωνία να κατατίζεται πριν να ξεκινάει προγραμματική περίοδος για να υπάρχει ο χρόνος επιλογής διαφόρων χρηματοστοτικών ενδιαμέσων εντός των σωστών πλαισίων και εντός της οικονομικής περίοδου. Μετά επιλογή των μεσαζόντων, των οικονομικών. Υπάρχει σύστημα βαθμολόγησης για την αξιολόγηση των υποψηφίων και θέλουμε να καθορίζονται ελάχιστε προδιαγραφέ και απαιτήσει για την επιλογή αυτών των μεσαζόντων. Χρειάζεται λεπτομέρεια όσον αφορά τον υπολογισμό των παραμέτρων που χρησιμοποιούνται για τι συμφωνίε σοφά τη εγγύηση. Τέταρτον, όσον αφορά παρακούση επιδόσεων και αναφορά. Συστήνουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δει κατά πόσο χρειάζονται καλύτεροι δείκτες επιδόσεων για καλύτερη παρακολούθηση των επιτευγμάτων του μέσου και το αν πετυχαίνει τα αποτελέσματα. Πέμπτη σύσταση. Επιτεύγματα του ΣΜΑΚ. Κυρίως τα δάνεια που δίδονται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δεν έχουν αρκετές εγγύησεις και καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εντοπίσαμε καθυστέρηση εκεί. Συστήνουμε λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο μέλλον να θέσει σαφέστερους στόχους που σχετίζονται καλύτερα με τους στόχους του μέσου. Και κατά τη διάρκεια του βίου του μέσου, ποια είναι η πρόοδος της επίστευξης των στόχων και πώς ελαχιστοποιείται το απόβαρο, αν θέλετε, τα εμπόδια, ούτω ώστε να δίδονται αποτελεσματικότερα οι πόροι της Ευρωπαϊκής Ενώσεως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με τα σωστά προγράμματα που αλλιώς δεν θα χρηματοδοτούνται. Τέλος Έκτη σύσταση. Το ελεκτικό συνέδριο επαναλαμβάνει ότι οι δαπάνες που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δικαιολογούνται από ωφέλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και να αποδεικνύεται ότι δεν θα μπορούσε αλλιώς να επιτευχθούν τα αδέοντα αποτελέσματα. Δηλαδή από υποστήριξε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Ότι δεν θα επιτυχαίναν αυτά τα αποτελέσματα με αποκλειστικά τοπική, περιφερειακή και εθνική χρηματοδότηση και πώς μπορούμε να γιστοποιήσουμε την προστιθέμενη αξία της Ευρωπαϊκή Ενώσεω με τη χρήση του μέσου. Η ειδική έκθεση συμπεριλαμβάνει και απαντήσει Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τα πορίσματά μα. Εμεί και υποφαινόμενο εκφράζουμε ικανοποίηση για τι περισσότερε συστάσει εκθέσει που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ρίχνοντα μια πρώτη ματιά στην πρόσφατη πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή για κανονισμό για την κατάρτιση του μελλοντικού προγράμματο για ανταγωνιστικότητα για τι επιχειρήσει και τι μικρομεσαίε επιχειρήσει, το COSME, για την επόμενη περίοδο 2014-2014, μάλλον 2014-2020, και το νομοθετικό πακέτο για το πρόγραμμα για τη χρηματοδότηση της έρευνας Horizon 2020 θεωρώ ότι πράγματι παίρνει τι συστάσει μα σοβαρά υπόψη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την δική έκθεση στην οποία αναφέρομαι. Κυρίω συστάσει που αφορούν του στόχου παρέμβαση, ε, δείκτε επιδόσεων, στόχου, ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία ε, και αυτό είναι ενθαρρυντικό για μένα. Κύριε Πρόεδρε, κυρίε και εξότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αυτό σημαίνει ότι ο έλεγχο τη αποτελεσματικότητα του μέσου ΣΜΑΚ ε, ήταν κάτι χρήσιμο και σχετικό και το ελεκτικό συνέδριο πιστεύει ειλικρινά ότι θα εξυπηρετήσει τους σκοπούς τους, θα χρησιμεύσει και στο Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια των συζητήσεων για μελλοντικά προγράμματα υποστηρίξεως των μικρομεσών επιχειρήσεων. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ κύριε Μπαλκό. Θα ήθελα να δώσω το λόγο τώρα στην εισηγήτρια. Κυρία Γκρέσλα έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ και ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαριστήσω το ηλεκτρικό συνέδριο. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η έκθεση γιατί μας λέει για πρώτη φορά κάτι για τα πιο σημαντικά ε, προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εγγυήσεις δηλαδή για τις ΜΜΕ. Είναι σημαντικό γιατί πραγματικά αφορά πάρα πολλέ επιχειρήσεις. Είναι ένα πρόγραμμα που ε, δρά σε μια σχέση 1 προς 10, μια πολλαπλησιαστική σχέση δηλαδή και είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί ήδη το 2009 βέβαια το ηλεκτρικό συνέδριο σύλλεξε αυτά τα στοιχεία και θα ήθελα να ρωτήσω αν εντωμεταξύ υπάρχουν και άλλα στοιχεία ίσως για κάποια αλλαγή της βασικής αυτής στάσης. Κατόπιν μου φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η κριτική του ηλεκτρικού συνεδρίου γιατί πραγματικά εδώ στο σώμα η μόνη μας ανησυχία είναι κατά πόσον είναι ορατή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είναι σαφές ότι δεν είναι πολύ ορατή με τα χρηματοδοτικά αυτά μέσα. Το επόμενο σημείο, η διαφάνεια. Αν σκεφτούμε πόσα δεν ξέρουμε για τα ε, χρηματοδοτικά μέσα, δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει τεράστια διαφάνεια αυτή τη στιγμή. Και το τρίτο είναι η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Επιτέλους θα έλεγα είναι σαφές το συνέδριο γιατί είπε ότι δεν απεδείχθη καμία ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Αυτό βέβαια είναι δραματικό γιατί εμείς θέλουμε να υπάρχει βέβαια μια ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και μια τέτοια έκθεση εμένα με σοκάρει γιατί βλέπω ότι πρόκειται για ένα μέτρο με πολύ τοπική εργασία δηλαδή ε, μικρές ε, επιχειρήσεις, ε, καταστήματα κλπ. Ωραία όλα αυτά και σημαντικά όλα αυτά. Αλλά δεν είναι δικό μας έργο και γι' αυτό εγώ στα συμπεράσματά μου είπα ξεκάθαρα ότι δεν είναι δικό μας έργο να συγχρηματοδομούμε συμπληρωματικά εθνικά προγράμματα ή να αντικαταστούμε εθνικά προγράμματα, αλλά ακριβώ αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή. Οι καινοτοπικές πτυχές θα έπρεπε να επιτυγχάνονται με μια τέτοια ευρωπαϊκή χρηματοδότηση απουσιάζουν. Δηλαδή εμείς αυτό που θα θέλαμε θα ήταν να χρηματοδοτήσουμε επιχειρήσεις οι οποίες είναι τόσο κεντρονοπικές που δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τράπεζες. Και κάτι τέτοιο δεν υπάρχει. Και μου φαίνεται ότι το σημείο αυτό αναφέρεται πολύ σημαντικά από το ηλεκτρικό συνέδριο στην έκθεσή του. Δηλαδή μέχρι εμείς δεν μπορέσαμε να χρηματοδότησει πολλά καινοτομικά ε, σχέδια και γι' αυτό εγώ έχω πολλές ερωτήσεις όσον αφορά τη χρηματοδότηση. Ο συνάδελφος Ρουιπίκ που ενδιαφέρεται για το πρόγραμμα ΣΥΚ ιδιαίτερα θα είχε αυτοκτονήσει φαντάζομαι το 2010 γιατί αποσύραμε πολλούς πόρους από το πρόγραμμα ΣΥΜ που δεν είχαν απορροφηθεί. 60 εκατομμύρια ευρώ σχεδόν μου φαίνονται πολλά και τίθεται το ερώτημα τώρα, έχει τη σωστή μορφή αυτό το πρόγραμμα. Το 2011 είχαμε πολύ λίγα χρήματα, α, ε, δανείσει, αλλά το 2010 πάρα πολλά. Θα πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε το θέμα του προγραμματισμού. Κατόπιν. ανέφερε ότι θα πρέπει να στραφούμε προς ένα θέμα που δεν έχει εξετάσει το ηλεκτρικό συνέδριο, δηλαδή το θέμα του κόστους διαχείρισης αυτού του μέσου. Ο συζητήτρια ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για το θέμα αυτό. Μπορεί κανένα να το δει μέσω των ε, στοιχείων, των λογιστικών στοιχείων των επιχειρήσεων νομίζω. Θα ήταν λοιπόν πάρα πολύ ενδιαφέρον να έχουμε τα στοιχεία αυτά προσπάθησα να λάβω υπόψη με τις επικρίσεις του ηλεκτρικού συνεδρίου και τις ε, εμπειρίες που έχω εγώ με χρηματοδοτικά μέσα. Και νομίζω ότι κάποια πρέπει να κάνει ακόμα η Κομισιόν και θα ήταν καλό να μάθουμε πότε θα, θα μας έρθει διαβασμένη η Κομισιόν. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ κυρία Κρέστρε. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Τόμας της Κομισιόν, Διευθυντή για την συνανισμό της χρηματοδότησης κλπ. Σας χαιρετίζουμε εδώ στην Επιτροπή και αναρωτιέμαι κατά πόσο μπορείτε να απαντήσετε στις ερωτήσεις της ηγήτριας. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εκπρόσωπε του Αλεκτικού Συνεδρίου, κυρία Γκρέσλε, πρώτα απ' όλα να σας πω ότι Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που συζητούμε αυτήν την έκθεση. Έχουμε συνεργαστεί πολύ στενά με το ελεγκτικό συνέδριο σε ό,τι αφορά αυτό το μηχανισμό εγγύσεων και έχουμε ανταλλάξει πολύ χρήσιμες ε, απόψεις. Όπως είπε και ο εκπρόσωπος του συνεδρίου, δεχτήκαμε τις περισσότερες συστάσεις. Τις λαμβάνουμε ήδη υπόψη και για την ε, προετοιμασία μας ε, και για το νέο κόσμο αλλά και για το Ορίζοντα 2020, πάρα πολύ επικοδομητική λοιπόν ε, και χρήσιμη ήταν ε, η ανταλλαγή αυτή απόψε, ένα εξωτερικό μάτι αν θέλετε που κοίταξε το πρόγραμμά μας, το σχεδιασμό του προγράμματός μας. Χαιρόμαστε επίσης που η εισηγήτρια πολύ ξεκάθαρα και αυτή λέει στο σχέδιο εκθεσή ότι πρόκειται για ένα από τα πλέον επιτυχημένα προγράμματα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Να απαντήσω σε κάποια συγκεκριμένα ερωτήματα. Ένα από αυτά ήταν ο συντελεστή μόχλευση. Αυτή τη στιγμή έχουμε ήδη φτάσει στα τέλη Σεπτεμβρίου 2011 το 15,8% συντελεστή μόχλευση σε σχέση με το 10%. Μάλλον με τα στοιχεία του 2010. Άρα 15,8 ευρώ ε, μακροχρόνιων εγγύσεων έχουμε χρηματοδοτήσει και όσο ε, προχωράμε μπορεί ο συντελεστής αυτός να αυξηθεί ακόμη περισσότερο σε συνάρτηση με τον όγκο και τον αριθμό μεσαζόντων. Ήδη λοιπόν έχουμε φτάσει στο 15,8% και δεν έχουμε φτάσει ακόμη στα ανώτατα όρια γιατί έχουμε και τη σύνταξη των νέων συμβάσεων και αύξηση του drawdown των νέων ε, των, των ήδη φυσταμένων συμβάσεων. Σε ό,τι αφορά τώρα τα τέλη και τις ε, αμοιβέ για το ΣΜΕΚ, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εγγύησεων, έχει ένα από τα χαμηλότερα ε, τέλη, τα οποία βασίζονται στην απόδοση, στις επιδόσεις και όχι τόσο στο κόστος. Συνολικά λοιπόν το ποσό των τελών είναι 6% σαν όριο. Το μέγιστο δηλαδή η διαχείριση του προγράμματος καλύπτει μία περίοδο 19 ετών, διότι μετά την περίοδο της δέσμευσης θα πρέπει να παρακολουθηθούν οι εγγύησει, τα δάνεια και αν υπάρχουν και ε, στάσεις πληρωμών από μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τέλος πάντων φτάνουμε στα 19 έτη και 6% ετήσια τέλη λοιπόν 0,32% κατά ανώτατο όριο για να απαντήσω στα πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα που ετέθησαν από την εισηγήτρια σε ό,τι αφορά και τη μόχλευση και τα τέλη. Δράτω με τις ευκαιρίες για να σας δώσω και κάποιες πληροφορίες ε, σε σχέση με τα loss rates, τους συντελεστές απώλειας. Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου του 2011, 23 εκατομμύρια είχαμε απώλειες από μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 6,8% περίπου δηλαδή των δημοσιονομικών μας δεσμεύσεων από τα 338 εκατομμύρια τα οποία είχαν δεσμευθεί. Είχαμε απώλειες στις τάξεις των 23 εκατομμύριων μέχρι στιγμής. Αυτά τα guarantee calls θα συνεχιστούν για καμιά δεκαετία ακόμη. Και επειδή είναι και πολύ δύσκολο όπως ξέρουμε, η κατάσταση οικονομική, ήταν το 11, θα είναι και το 12, ίσως να υπάρξουν και άλλες απώλειες άρα να αυξηθεί αυτό το ποσοστό. Πάντως τα κονδύλια τα οποία έχουν διατεθεί ή δεσμευθεί νομίζω ότι θα είναι πάνω από επαρκή. Να τα υπόψη και το νοτατόριο. όριο. Αυτές είναι οι απαντήσεις που έχω να δώσω στα συγκεκριμένα ερωτήματα και φυσικά αν θέλετε και πρόσθετες πληροφορίες είμαι στη διάθεσή σας. Ό,τι αφορά τα σημεία και τις συστάσεις ε, του ελεκτικού συνεδρίου και της εισηγήτριας, νομίζω ότι θέτουν δύο σημαντικά ζητήματα. Την αιτιολόγηση αφενός της λογικής παρέμβασης και αφετέρου την επίδειξη αν υπάρχει προσθέμενη ευρωπαϊκή αξία. Ήδη έχουμε λάβει υπόψη στο σχεδιασμό του νέου προγράμματος ε, τα δύο αυτά στοιχεία. Πράγματι, Όταν σχεδιάστηκε το πρόγραμμα, δηλαδή το 2007, οι βασικοί στόχοι του προγράμματος είχαν υποδιαιρεθεί. θέμενη ευρωπαϊκή αξία, όπως τότε είχαμε τεκμηριώσει, ήταν διαφορετικά τα κριτήρια, είχαμε και κάποια στόχους γεωγραφικής κάλυψης, έχουμε φτάσει ε, σε 19 διάμεσες χώρες ορισμός λοιπόν ε, της ε, προσθέμενης ευρωπαϊκής αξίας ενδιαφέρει σε σχέση με αυτό που χρησιμοποιεί η συγγήτρια. Δεχτήκαμε τις συστάσεις και θα ακολουθήσουμε την άποψη αυτή. Και θα αντιλαμβανόμαστε πλέον, θα ορίζουμε λίγο διαφορετικά την ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία και για το ε, κόσμο και για το Horizon 2020. Το έχουμε λάβει υπόψη μα και στι μελέτε αντικτύπου. Ο συνάδελφο από την επιχείρηση επιχειρήσει ίσω θα προσθέσει κάτι πάνω σε αυτό. Έπειτα, ειδική σύσταση, το ανέφερε και το συνέδριο, για την επιλογή των χρηματοοικονομικών μεσαζόντων. Σύστημα βαθμολόγηση. Μέχρι στιγμής και δεν νομίζω το αμφισβητεί το συνέδριο, η ανεξάρτητη αξιολόγηση, δηλαδή δεν αμφισβητεί ότι είχαμε μια καλή επιλογή μεσαζόντων. Και ίσως και για το μέλλον θα πρέπει απλά να το τεκμηρώνουμε καλύτερα. Αλλά νομίζω ότι στην φάση αυτή με 19, συγγνώμη, με 3, όχι 19, με 31 μεσάζοντες, βλέπουμε περισσότερο να δρομολογούν νέα προϊόντα. Άρα νομίζω ότι κοιτάοντας ε, ε, προς τα πίσω δεν νομίζω ότι θα είχαμε διαφορετικά αποτελέσματα με ένα σύστημα βαθμολόγησης. Οι συστάσεις σας πάντως θα ληφθούν υπόψη και θα το δούμε και όσο θα εξελίσσεται το πρόγραμμα. Ένα τελευταίο θέμα είναι νομίζω η χρηματοδότηση της καινοτομίας. Έχουμε διατυπώσει προτάσεις για δύο προγράμματα, το COSME και για το ορίζοντα 2020. Διαφορετική θα είναι η εστίαση, θα επικεντρωθούμε στην καινοτομία και σε άλλες πτυχές. Μεταξύ των δύο μέσων αυτών και εργαλείων νομίζω ότι θα μπορέσουμε στο μέλλον να εστιάσουμε καλύτερα στα μέσα τα οποία ε, έχουν να κάνουν πιο αποκλειστικά με την καινοτομία και, ε, πια και ποια όχι. Το ΣΜΕΓ σίγουρα δεν είναι ένα εργαλείο που καταρχήν είχε ως αποκλειστικό του στόχο την καινοτομία. Θα δούμε λοιπόν ότι κάποιες μόνο μικρομεσαίες επιχείρησεις και όχι όλες επωφελήθηκαν από το πρόγραμμα γιατί δεν έχουν όλες ε, το σκέλος της καινοτομία στο πρόγραμμά τους. Άρα και σε αυτό αλλά και στα μελλοντικά προγράμματα θα πρέπει να υπάρχει ένα πιο στοχευμένο προς την καινοτομία πρόγραμμα. Θα σταματήσω εδώ και θα απαντήσω στα ερωτήματά σας εφόσον ε, έχετε να μου θέσετε. Επιπλέον ερωτήματα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Τόμας. Ναι, έχουν ζητήσει και άλλους ε, λόγο. Καταρχήν η ψυχήτρια και μετά η κυρία Ιβάνω και η κυρία Κιτσέσκοβα. Η κυρία Γκρέσλε πρώτα. Εγώ είχα ρωτήσει και πόσες αιτήσει έχουν απορριφθεί. Έχετε κάτι να μας πείτε αυτό, πάνω σε αυτό. Και επίσης αυτά τα 23 εκατομμύρια ευρώ απολειών πάνω σε ποιο αριθμό βάσης στηρίζονται. Ευχαριστώ, Ρε Πρόεδρος. Να συλλέξουμε λιγάκι τις ερωτήσεις. Η συνάδελφος Ιβάνοβα έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα πραγματικά να σας πω ότι χαιρετίζω την ειδική αυτή έκθεση του ηλεκτρικού συνεδρίου για το μέσο ΣΜΕΚ. Και είμαι ιδιαίτερα ευτυχής γι' αυτό γιατί θεωρώ ότι αυτή η έκθεση δίνει πάρα πάρα πολύ χρήσιμα στοιχεία για την εργασία μας στην Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού. Ιδίω στη δική μου εργασία για την ε, ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για το 2010. Αυτή είναι μία από τις λίγες εκθέσεις ε, του ελεκτικού συνεδρίου που μπορεί να με βοηθήσει στα δικά μου έγγραφα και θεωρώ ότι πολλά από τα συμπεράσματα του συνεδρίου που αναφέρθηκαν από το πρόσωπο του συνεδρίου όσον αφορά τα μεσάζοντα στοιχεία, την έλλειψη των ε, δικτών για την προστιθέμενη αξία κλπ. Θέλω να ρωτήσω το συνέδριο, προβλέπετε να δώσετε μια συνοχή για την εξτάση ποια είναι η πρόοδος που επιτεχάνετε, ποια είναι η συνέχεια που δίνετε στις συστάσεις σας και επίσης προβλέπεται ίσως κάποια ειδική έκθεση για τα, οικονομικά, για τα μέσα συγγνώμη, ε, οικονομικής ε, μηχανικής financial engineering και αν ναι πότε προτίθεστε να υποβάλλετε μια τέτοια έκθεση. Σας ευχαριστώ κύριε Ιβάνοβα. Η κυρία Τσέσκοβα έχει το λόγο. Εκτός μικροφώνου. Σας ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Ε, θεωρώ πάρα πολύ σε αυτή την έκθεση. Πριν να ε, έρθω στο κοινοβούλιο, εργαζόμουν πάρα πολύ συχνά με μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Τσεχία και γι' αυτό θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που μας δίνετε μία εικόνα του μηχανισμού αυτού τώρα και επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω την Κομισιόν η οποία προέβλεψε υποστηρίξη των μηνεύσεων στον τομέα αυτό. Ε, δύο θέματα με ενδιαφέρουν εμένα ιδιαίτερα όσον αφορά τα συμπεράσματα του ελεκτικού συνεδρίου. Το πρώτο είναι ότι αυτό το πρόγραμμα θα πρέπει να συγκεντρωθεί περισσότερο στις ε, επενδύσεις αλλά και στην επαναχρηματοδότηση του χρέους. Δεν ξέρω, μπορούμε να έχουμε κάποια στοιχεία να αφορά αυτή τη δυνατότητα, δηλαδή τη χρηματοδότηση χρέους. Και το δεύτερο που θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό και ενδιαφέρον είναι ο τρόπος με τον οποίο ε, καταμετρούνται οι επιπτώσεις αυτού του σχεδίου. Γιατί στην έκθεση του ηλεκτρικού συνεδρίου υπάρχει ένα αποτέλεσμα που αφορά τον αριθμό των θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν λόγω της υποστήριξης αυτής. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η δημιουργία θέσεων απασχόλησης είναι ένας από τους στόχους του χρηματοδοτικού αυτού μέσου. Και αναφέρεται δωρητά ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει σαφής αξιολόγηση των εν λόγω επιπτώσεων. Γιατί αναφέρεται μόνο ο αριθμός ε, των θέσεων απασχόλησης εν λόγω εταιρείας, χωρίς να αναφέρεται ο αριθμός των θέσεων απασχόλησης που δημιουργήθηκαν λόγω της χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά είναι τα στοιχεία που με ενδιαφέρουν και θα ήθελα να ακούσω τις απαντήσεις σας, αν έχετε να μας πείτε κάτι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Τσέσκοβα. Συνάδελφο Ρούβικο, τελευταίο τελευταίος σε αυτό το γύρο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι αυτή η χρηματοδότηση των ΜΜΕ ακριβώς στη σημερινή κατάσταση της κρίσης και της κρίσης χρηματοδότησης ιδίως των ΜΜΕ καταδεικνύει πόσο σημαντικό είναι κάτι τέτοιο και θα ήθελα απόλυτα να υποστηρίζω την κυρία Γκρέσλε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, θα πρέπει να ασχολείται με ανεξάρτητα μέσα και όχι να προωθήσει μια συγχρηματοδότηση η οποία έχει διαφορετικούς στόχους και η οποία βέβαια οδηγεί και σε έναν αναγνωσμό με τις εθνικές και περιφερειακές τράπεζες. Γιατί μια τράπεζα εθνική σκέφτεται πού μπορεί να έχει το καλύτερο όφελος και κατά τη γνώμη μου προσφέρει στις ΜΜΕ ε, πρέπει να προσφέρουμε εμείς εδώ ε, χρηματοδότηση όταν δεν μπορεί να γίνει μέσω της τράπεζας. Τι σκοπεύει λοιπόν η Κομισιό να κάνει για να μπορέσει να εξαλείψει τον ανομισμό που έχει με τις εθνικές και περιφερειακές τράπεζες και πώς θα μπορέσει αυτή την προσφορά της να την καταστήσει πιο ελκυστική. Να μην είναι δηλαδή μόνο ένα σχέδιο τελικά ενίσχυση των τραπεζών. Θα σε ευχαριστώ πολύ κύριε Ρούμπιχ. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Τόμας της Κομισιόν για να απαντήσει στις ερωτήσεις αυτές. Έχετε το λόγο κύριε Τόμας. Σας ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα για να δώσω στην κυρία Γκρέσλε τι απαντήσει Τα 23 εκατομμύρια τα οποία ανέφερα ήταν κάποιες κλήσεις ε, της τράπεζας προς την Κομισιόν για τις εγγύησεις. Πρόκειτο δηλαδή για κάποιες μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες είχαν πρόβλημα επιτόπου. Είναι στοιχεία από μέχρι το Σεπτέμβριο του 2011 και μπορούμε να σας δώσουμε σε όλα τα στοιχεία, κυρία Γκρέσλε, για να έχετε όλα τα στοιχεία στη διάθεσή σας. Ό,τι αφορά τις απορριφθήσεις ε, αιτήσει, να σας πω ότι εμείς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρεμβαίνουμε με βάση προτάσεις που διατυπώνει το EIF. Μία αίτηση έχουμε απορρίψει μέχρι στιγμής όπως αναγνωρίζει και το συνέδριο, έχουμε αναπτύξει ένα ε, μάλλον πλήρη συστήματα για την επιλογή των δημοσιολαβητών, των μεσαζόντων. Αυτή τη στιγμή όμως, σήμερα δεν μπορώ να σας πω συγκεκριμένα τις απορρίψεις που έγιναν ε, την, σε επίπεδο EIF. Πόσες αιτήσει έλαβε και πόσες απέρριψε στην πρώτη φάση της επιλογής. Εμείς ε, στο δεύτερο στάδιο μία αίτηση, όπως σας είπα, έχουμε απορρίψει. Κάποιες άλλες ε, ερωτήσεις τώρα να απαντήσω. Πρώτα απ' όλα, η κυρία Ιβάνοβα, γιατί ο follow-up που θα έχει το συνέδριο θα απαντήσει φαντάζομαι το συνέδριο σε αυτό το ερώτημα, αλλά να σας πω ότι εμείς τουλάχιστον από τη δική μας πλευρά Ήδη έχουμε δείξει με τα δύο προγράμματα Κόσμο και Ορίζον 2020 της τη αξιολόγηση των επιπτώσεων. Έχουμε δείξει ότι θα λάβουμε πολύ σοβαρή υπόψη μας τι συστάσεις του Ελληνικού Συνεδρίου. Σε ό,τι αφορά τον ανταγωνισμό, την περιφερειακέ Τράπεζε και πάλι σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Προστέμενη Αξία και το ζήτημα το οποίο έθεσε η κυρία Τσέσκοβα για την αναχρηματοδότηση του χρέους. Για τα θέματα αυτά βλέπουμε ότι είναι πολύ λεπτή η επιτευχή της ισορροπίας. Στόχος της χρηματοδότησης, σε σχέση με το στόχο της χρηματοδότησης, από την ανάλυση φαίνεται ότι σε κάποιες περιπτώσεις έχουμε χρηματοδότηση αμυγός της καινοτομίας, ενώ σε άλλες περιπτώσεις έχουμε αναχρηματοδότηση και working capital financing. Κάποιοι αυτό το ε, επικρίνουν. Αν δεν κανείς όμως την ανεξάρτητη αξιολόγηση, κάτι το θεωρούν πλεονέκτημα. Ε, financing ή working capital financing, δηλαδή για μικρή χρονική περίοδο λόγω της κρίσης. Είναι ένα θέμα συζήτησης αυτό. Θα το διευκρινίσουμε στο μέλλον. Αλλά για την ανεξάρτητη αξιολόγηση αυτό θεωρήθηκε πλεονέκτημα. Δηλαδή, εν καιρό ε, δύσκο, ε, κρίσης οικονομικής να μπορεί να γίνει αυτή ένα αναχρηματοδότηση. Είναι θετικό. It is, ε, Κάποιες άλλες ε, φορές όμως φάνηκε ότι αυτό συνιστά μη επαρκή προστέμενη αξία. βλέπουμε να υπάρχει μια αντίφαση σε ό,τι αφορά τι περιφερειακέ τράπεζε. Βλέποντα το μηχανισμό εγγύησεων επιχειρήσεων τώρα, όπω έχει αυτό ο μηχανισμό και τι θα σα πω για το μέλλον. Όσο έχει αυτή τη στιγμή αυτό ο μηχανισμό. θα έλεγα ότι στι περισσότερε περιπτώσει είναι πολύ μικρό για να ανταγωνιστεί κάποια εθνικά προγράμματα και μηχανισμού. Γι' αυτό λοιπόν είναι και δικαιολογημένο το ότι ψάχνουμε την ευρωπαϊκή προστέμενη αξία και όχι να είμαστε ανταγωνιστικοί προς καθαρά εθνικά σχέδια. Προχωρώντας τώρα στη νέα δημοσιονομική περίοδο, αλλά βέβαια και με την επιφύλαξη των αποφάσεων που θα λάβουν ε, οι αρχές ε, για τον προϋπολογισμό και σε σχέση και με το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Και για το κόσμο και το ορίζον 2020, αλλά και στις προτάσεις για ένα νέο μέσο τομέα των εξωτερικών ταμείων, η Κομισιόν έχει μια διαφορετική κλίμακα ε, προγραμμάτων να προτείνει. Και σε επίπεδο εθνικών ταμείων και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικώ. Ε, έχουμε και συγχρηματοδότηση με εθνικά μέσα στον τομέα της διαθροτικής χρηματοδότησης. Θα ακολουθήσουμε μια νέα προσέγγιση για να υπάρχει συμπληρωματικότητα και να μην υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ περιφερειακών μηχανισμών συγχρηματοδότησης και ευρωπαϊκής χρηματοδότησης. Θέλουμε να υπάρχει συμπληρωματικότητα. Αυτό είναι ο στόχος μας. Ήμουν παρόν και στις προηγούμενες συζητήσεις. Πρέπει να σας πω ότι η συμπληρωματικότητα αυτή θα πρέπει να εξασφαλιστεί και μέσω της απλούστευσης θα πρέπει να λέμε υπόψη μα τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Δεν πρέπει να δημιουργήσουμε για αυτέ ένα ιδιαίτερα πολύπλοκο περιβάλλον και να μπορούν, ε, θα πρέπει εύκολα να μπορούν να διακρίνουν μεταξύ των διαφορών επιπέδων ευρωπαϊκού, εθνικού, περιφερειακού. Πρέπει να υπάρχει επίση και μεγαλύτερη ορατότητα και για του τελικού δικαιούχου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπορείτε να πείτε και κάτι συμπληρωματικά για κάτι που εθίγει στην, στο πρώτο γύρο από την ίδια την εισηγήτρια. Το θέμα της προσθέμενης αξίας δηλαδή. Ακούσαμε τη σχετική επίκριση του ηλεκτρικού συνεδρίου εσείς τι έχετε να πείτε από αυτού ή υπάρχει και κάποια σκέψη στο μέλλον να αυξηθεί αυτή η ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία με μια αλλαγή του κανονισμού για τη χρηματοδότηση των ΜΜΕ. Äh, λοιπόν, μήπως μπορείτε ίσως να απαντήσετε στο σημείο αυτό που εθίγει από την εισηγήτρια στο πρώτο γύρο, αλλά από ξέρω δεν έχει απαντηθεί αλλά είναι σημαντικό για όλοι μας στην Επιτροπή. Πώς μπορείτε κάτι να πείτε από αυτού. Δεν έχω να πω τόσα πολλά όσον αφορά το θέμα του ΦΠΑ. Φοβούμαι ότι δεν είναι κάτι στο οποίο μπορώ να υπησέλθω σε λεπτομέρειες. Προσπαθούμε, όπως είπα, μέσω του σχεδιασμού του μέσου θα προσπαθήσουμε να εξασφαλίσουμε ότι η νέα προστιθέμενη αξία θα υπάρξει στο μέλλον. Όσον αφορά το ΦΠΑ, προτιμώ να μην μπω στα εδάφη, στα χωράφια άλλων υπηρεσιών. Προέδρο πρόεδρος εκτός μικροφώνου. Ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Μπορείτε να μας δώσετε γραπτός ενδεχομένως κάποιες πληροφορίες, αν έχετε δυνατότητα. Απάντηση βεβαίως, όσον αφορά την προστιθέμενη αξία την ευρωπαϊκή, στην αξιολόγηση αντικτύπου για το νέο μέσο, για τα νέα μέσα το αναφέρουμε, να είναι ξεκάθαρο. Προσπαθήσαμε, λαμβάνουμε όπως τι τάσει του ελεκτικού συνεδρίου όσον αφορά τους δείκτες συνεπιών, εν αντιθέσει με τους νέους δείκτες εκρών, και αυτό είναι μέσω του σχεδιασμού του αντιμετωπίσμα. Όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα του ΦΠΑ, από ό,τι κατάλαβα, εκεί δεν μπορώ να σα δώσω πληροφορίε. Θα, προσπαθώ, θα προσπαθήσω να το διαβάσω στις αρμόδιες υπηρεσίες. Ευχαριστώ. Now, πριν μπούμε στον τελευταίο γύρο, ο κύριος Μπάλκο και μετά ο λόγος θα δοθεί στην κυρία Γκρέσλε. Πρώτα ο κύριος Μπάλκο έχει το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως και η κυρία Ιβάνα Πανιτσεύσκο. Θα ήθελα να απαντήσω στην κυρία Ιβάνοβα μάλλον. Εδώ διερωτήθηκε για τη συνέχεια. ο έλεγχος για το μέσο αυτό του οικονομικού μηχα... μηχανικής αντιμετώπισης, financial engineering, ε, είναι με έκθεση δημοσιευθεί σύντομα. Θα αφορά το 2012 και δημοσιευθεί πάρα πολύ σύντομα. Σήμερα ε, ε, λάβαμε email από συναδέλφους και λένε ότι έχει εγκριθεί. Εστιάζεται και επί και αποδοτικότητας αυτό των μέσων χρηματοστικής οικονομικής, μηχανικής μάλλον, και πρώτα απ' όλα για την ποιότητα της αξιολόγησης της χρηματοδοτήσεως μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ποιο είναι το κατάλληλο πλαίσιο για τη χρήση των μέσων και τι γίνεται με την αποτελεσμάτων. Ενδιαφέρεται ο φορέας μας για αυτό το θέμα. Και σε κάνα δύο χρόνια θα εξετάσουμε ποια θα είναι η συνέχεια που θα δοθεί. Λοιπόν, θα συνεχίσω στη μητρική μου γλώσσα, στα σλοβακικά. Θα ήθελα να πω ότι εξετάσαμε τα διάφορα προβλήματα που υπάρχουν špecifickej A my práve v tomto bode iba poukazujeme na problém, ktorý je s merateľnosťou počtu vytvorených pracovných miest a na Υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα για την ώρα. συγγνώμη πλευρά Υπάρχει ένα πρόβλημα αφορά την γλώσσα που χρησιμοποιείται τώρα. Thank you. This was my answer on questions. Και αυτή ήταν η απάντησή μου, λέει ο μιλητής. So If there was no translation... Αν δεν υπήρξε, δεν λειτουργήσε, υπήρχε τεχνικό πρόβλημα, μπορώ να το απαντήσω. Ναι, υπήρχε πρόβλημα, λέει ο πρόεδρος, πράγματι. Ναι, υπάρχει πρόβλημα. Την πρώτη φορά δεν υπήρξε, δεν πέρασε το μήνυμα. Υπήρχε τεχνικό πρόβλημα, όπως σας είπαμε από ελληνική καμπίνα. Μπορεί Μήπως μπορείτε το πρώτο τμήμα της απάντησής να το απαντήσετε. Α, ναι, ναι, ναι, ναι. ευχαριστώ. ευχαριστώ. I explain, I explain in English. Θα εξηγήσω αγγλιστή. Η κυρία Τσέσκοβα έθεσα ένα ερώτημα. Αριθμό θέσεων εργασίας. Αυτό αναφέρεται στην παράγραφο 68 της εκθέσεως. Εδώ, στην 68, αναφέρουμε ένα πρόβλημα που διαπιστώσαμε στον έλεγχο επιδόσεων. Αναφέρουμε ότι είναι δύσκολο να μετρήσουμε τον αριθμό θέσεων που δημιουργείται, που δημιουργούνται μάλλον και κάναμε και τις κατάλληλες συστάσεις για να βελτιωθεί αυτό. Ευχαριστώ κύριε Μπάλκο, λέει πρόεδρος. Για να ολοκληρώσουμε σημαίνει με συζήτηση, θα ήθελα να δώσω το λόγο στην εισηγήτρια. Κύριε Γκρέσλε, θα ήθελα να ξαναρωτήσω την Κομισιόν όσον αφορά το διοικητικό κρόστος. Αυτό το 6%. Εδώ μεταξύ μας μπορώ να σας πω που μου φαίνεται υπερβολικά 6% γιατί το 7% είναι αυτό που παίρνουν τεράστια δίκτυα για διαχείριση των δικτύων αυτών. 6% μου φαίνεται λοιπόν εδώ πολύ. Θα με ενδιαφέρει να δω κάποια συγκριτικά στοιχεία. Αλλιώς, ε, πολύ, πολύ <laughs> καρποφόρο είναι αυτή η υπόθεση. Λοιπόν, πώς το υπολογίζετε αυτό. Κατά τα άλλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για όλα όσα μας είπατε και περιμένουμε τα στοιχεία που θα μας δώσετε ακόμα. Πρόεδρος, ευχαριστώ κυρία Γκρέσλε. Μπορείτε για το διοικητικό κόστος ήδη τώρα να μας πείτε κάτι κύριε Τόμας ή θέλετε να μας το δώσετε γραπτά. Μπορούμε να στείλουμε γραπτός. Όπως σας είπα 6% κατά τη διάρκεια ζωής του προγράμματος. Πάνω από 19 χρόνια. 0,32% ανά έτος το χαμηλότερο κόστος διαχείρισης ιουδήποτε προγράμματος και ιονδήποτε μέσων, μέσου. Θα σας στείλουμε λεπτομέρειες. Είναι 0,32% ανά 6% κατά τη διάρκεια ζωής του προγράμματος μέχρι ότου εκπνεύσει τελευταία εγγύηση. Και μέχρι τόσο καταβληθούν τα ποσά, δηλαδή 19 ετής περίοδος, 19 χρόνια. Ευχαριστώ κύριε Γκρέσλερ αλλά δεν ε, χρειάζεται να εργαστείτε κάθε χρόνο, δεν ασχολείστε κάθε χρόνο, δίνετε τα χρήματα και μετά συνεχίζει το πράγμα, ξέρω εγώ, 7-8 χρόνια. Λοιπόν, μήπως έχει καμιά φορά υπολογιστεί δύο φορές το κόστος. Πρόεδρος, κοιτάξτε, ίσως πραγματικά χρειάζεται να πάρουμε κάποιες συμπληρωματικές ε, λεπτομερείς πληροφορίες ε, εδώ στην Επιτροπή μας για να καταλάβουμε καλύτερα κατά πόσο το ποσό αυτό είναι ε, υπερβολικά υψηλό ή υπερβολικά χαμηλό. Θα σας ήμουν να μα δίνετε τα στοιχεία αυτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Τόμα για το σημείο αυτό και ιδίω τον... ευχαριστώ τον κύριο Μπάλκο και θα ήθελα να κλείσουμε αυτό το σημείο της σημερινής διάταξης και να περάσουμε στο σημείο 7 θα ήθελα να χαιρετήσω εδώ την κυρία Τετέσσα Σανταλόβα του Ελεκτρικού Συνεδρίου. Η συγκίση είναι ο κύριο Μπαρτιθάση και Σανταλόβα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια για την εκλογή σα και τη κυρία Σιβάνοβα, Είμαι πολύ ευχαριστημένη. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, εξεταμένοι του Κοινοβουλίου, κυρίε και κύριοι, σα παρακαλώ επιτρέψτε μου να παρουσιάσω την ειδική έκθεση όσον αφορά τι διαδικασίε επιτροπή να ασφαλιστεί η αποτελεσματική διαχείριση του ελέγχου των κρατικών ισχύσεων. Θα ήθελα να σας ε, εξηγήσω λίγο τι θα πει ε, κρατική ενίσχυση και ποιες είναι οι διαδικασίες ελέγχου. Οι κρατικές ενισχύσεις ορίζονται στο 107 τις συνθήκες για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως οποιαδήποτε ενίσχυση δίδεται από ένα κράτος μέλος ή από κρατικού πόρους υπό οποιοδήποτε μορφή που στρεβλώνει ή απειλεί να στρεβλώσει τον ανταγωνισμό ευνοώντας ορισμένες επιχειρήσεις ή παραγωγή ορισμένων αγαθών στον βαθμό που αφορά το εμπόριο μεταξύ κρατών μελών. Επομένω, οι επιδοτήσει οι οποίε δίδονται είτε σε ιδιώτε ή τα γενικά μέτρα τα οποία ε, είναι ανοιχτά για όλε τι επιχειρήσει, γενικά δεν συνιστούν κρατική ενίσχυση. Οι κρατικέ ενισχύσει ε, παρέχονται με διαφορετικού τρόπου. Η πιο συχνή μέθοδο είναι οι επιδοτήσει ή φοροαπαλλαγέ. Άλλε μορφέ είναι τα λεγόμενα μαλακά δάνεια, εγγυήσει, προτιμησιακή φορολογική μεταχείριση ή συμμετοχή ε, από τα κράτος ε, στο κεφάλαιο. Οι κρατικέ ενισχύσει μπορούν να παρέχονται από την εθνική, την ομοσπονδική, την περιφερειακή, την τοπική κυβέρνηση, αλλά και από κρατική κρατικούς φορείς. Ευθύνη για τον αποτελεσματικό έλεγχο των κρατικών νησιών, την έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συγκεκριμένα η ΓΔ Ανταγωνισμός, που είναι και αρμόδια για τον έλεγχο των κρατικών νησιών σε όλους τους οικονομικούς τομείς εκτός από τη Γεωργία και την Αλία. Στόχος ε, του ελέγχου της Κομισιόν για τις Κρατικές Ενισχύσεις είναι να διασφαλίσει ότι οι κρατικές ενισχύσεις ε, που δίνονται από τα κράτη-μέλη είναι συμβατές με την εσωτερική αγορά, Άρα να εξασφαλιστεί ότι οι κρατικέ παρεμβάσει δεν στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό και το εμπόριο εντό Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν πρέπει να κοινοποιούν στην Κομισιόν όλα τα σχέδια ε, για μέτρα κρατικών ενισχύσεων και πριν τα εφαρμόσουν να έχουν την έγκριση τη Κομισιόν, που είναι η μόνη αρχή η οποία μπορεί να θεωρήσει και να κηρύξει ένα μέτρο κρατική ενίσχυση συμβατό με τη συνθήκη. Έχει λοιπόν ε, πάρα πολύ μεγάλη διακριτική ευχέρεια στον τομέα αυτό. Εάν το μέτρο το οποίο ε, έχει ζητηθεί ε, αποτελεί ε, κρατική ενίσχυση και θεωρείται συμβατό από την Κομισιόν, συμβατό με την Αστική Αγορά, τότε εγκρίνεται. Αν όμως η Κομισιόν αμφιβάλλει για το κατά πόσον υπάρχει συμβατότητα με την αγορά, θα ξεκινήσει τη διαδικασία της επίσημης έρευνας, Formal Investigation Procedure, βάσει των πληροφοριών που θα λάβει και την ανάλυση που θα πραγματοποιήσει, λαμβάνει τελική απόφαση. Όλοι οι φορεί τη ιστορική αγορά ή άλλοι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα να κάνουν καταγγελία στην Κομισιόν αν πιστεύουν ότι έχουν επηρεαστεί αρνητικά από μια ενίσχυση που έδωσε ένα κράτο μέλο και η οποία ε, στρεβλώνει ή απειλεί να στρεβλώσει τον ανταγωνισμό. Οι καταγγελίε αναλύονται, ερευνώνται από την Κομισιόν στο πλαίσιο τη λεγόμενη διαδικασία καταγγελία, complaint procedure. Επίση, μπορεί η Κομισιόν να ε, πάρει πρωτοβουλία, να δρομολογήσει δική της έρευνα για την συμβατότητα οποιαδήποτε, οποιασδήποτε ενίσχυσης με βάση τις ε, πληροφορίες που είναι ε, ευρύτερα. Κάποια στοιχεία τώρα για τις ε, διαδικασίες ελέγχου που ακολουθούμε. Στόχος μας πρώτα απ' όλα είναι να αποτιμήσουμε το κατά πόσον είναι αποτελεσματική διαχείριση του ελέγχου της ε, κρατικής ενίσχυσης. Επικεντρωνόμαστε πρώτα απ' όλα στα συστήματα κοινοποιήσεων, ε, της διαχείρισης των καταγγελιών. Μετά βλέπουμε κατά πόσον ε, η Κομισιόν έχει δομές, επαρκείς δομές διαχείρισης για να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις υποθέσεις κρατικών ενισχυσόντας των προθεσμιών. Τρίτον, πρέπει να δούμε κατά πόσον παρακολουθεί η Κομισιόν τον αντίκτυπο του ελέγχου κρατικών ενισχύσεων. Το, για την περίοδο 2008-2010 ήταν η περίοδος που καλύφθηκε Είδαμε την ε, οργάνωση, τη διαδικασία λήψης αποφάσεων ε, και τις διαδικασίες παρακολούθησης Κομισιόν, αλλά δεν έχουμε ε, αξιολογήσει το κατά πόσον ήταν ορθές οι αποφάσεις της Κομισιόν και καλύψαμε τους τομείς για τους οποίους είναι αρμόδια γάμα δέλτα ανταγωνισμού. Πρόκειται για το 96% όλων των κρατικών ενισχύσεων που χορηγήθηκαν το 2009 χωρίς τους σιδηροδρόμους. Εξετάσαμε περίπου 50 προκοινοποίησεις, 30 καταγγελίες, 40 υποθέσεις παρακολούθησης και 10 υποθέσεις ανάκτησης. Είχαμε συνεντεύξεις με το προσωπικό που ήταν αρμόδιο για την διαχείριση αυτών των υποθέσεων, καθώς και με διευθυντές 10 διαφορετικών μονάδων της ΓΔ ανταγωνισμού. Και εξετάσαμε τα σχετικά έγγραφα, κάναμε και αναλυτικές δοκιμασίες. Επισκεφθήκαμε 8 κράτη-μέλη. Συλλέξαμε επιπλέον επιπρόσθετες πληροφορίες από 44 κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς για το κατά πόσο αντιλαμβάνονται και πώς εκτιμούν τις διαδικασίες της Κομισιό χρησιμοποίησαμε τις απόψεις τους μόνο εάν ήταν σύμφωνοι και μια μεγάλη πλειοψηφία άλλων εμπλεκομένων φορέων. Να σας δώσω τώρα κάποια αποτελέσματα. Ένα από, το βασικό, από τα βασικά μηνύματα που προέκυψαν ήταν ότι δεν έχει επαρκείς διασφαλίσεις η Κομισιόν ότι καλύπτει και ε, ασχολείται με όλες τις σχετικές υποθέσεις ε, κρατικής ενίσχυσης και γι' αυτό λάβαμε κάποια μέτρα για να βελτιώσουμε τη συνεργασία μας με τα κράτη-μέλη σε ό,τι αφορά την, ε, την υποχρέωση κοινοποίηση που έχουν. Δεν ήταν επαρκή αυτά τα βήματα όμως. Κυρίως βασιζόμαστε σε καταγγελίες από τρίτους για να δούμε κατά πόσον δεν έχουν κοινοποιηθεί κάποιες κρατικές ενισχύσεις. Υπάρχουν περιθώρια λοιπόν για να ε, κάνουμε πιο συχνή χρήση των ερευνών από ίδια πρωτοβουλία. Από νομικής πλευράς δεν μπορεί όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συστηματικά να παρακολουθεί και να αξιολογεί την ε, αξιοπιστία των διαδικασιών που ακολουθούν τα κράτη-μέλη. Είναι περιορισμένες οι δραστηριότητες παρακολούθησης. Άρα υπάρχει κίνδυνος να υπάρχουν ε, κρατικές ενισχύσεις τις οποίες δεν ε, μπορούμε να ανοιχνεύσουμε. Ένα άλλο σαφές μήνυμα είναι ότι είναι χρονοβόρες οι διαδικασίες σε επίπεδο επιτροπής και δεν υπάρχει επαρκής διαφάνεια. Πολλά από τα στοιχεία και φάσεις ε, μπορούμε να πούμε ότι έχουν καλή διαχείριση και καλή οργάνωση, αλλά πολλές φορές χρειάζεται πολύ χρόνο μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Επίσης έχουν αυξηθεί οι καταγγελίες, άρα έχουμε καθυστέρηση ε, χρονική και δεν λαμβάνουν ε, οι φορείς ε, επαρκείς πληροφορίες για την πρόοδο της αντιμετώπισης των, και επεξεργασίας των καταγγελιών τους. Άρα μικρή διαφάνεια είναι το αποτέλεσμα. Τρίτο βασικό μήνυμα. Δεν αξιολογείται από την Κομισιόν ο εκ αντίκτυπος του ελέγχου της κρατικής ενίσχυσης συνολικά δεν υπάρχουν αξιόπιστα στοιχεία. Αυτό παρακολεί τις προσπάθειες Κομισιόν. Έχουμε ένα πίνακα ε, βαθμολογίας, ε, το scoreboard, το οποίο όμως έχει πολλά, ε, πολλές ελλείψεις. Αυτό όμως είναι το βασικό εργαλείο αναφορών που έχουμε. έλλειψη πληρότητας και παρκούς αξιοπιστίας και συγκρισιμότητας. Έρχονται αρκετά καθυστερημένα τα στοιχεία. Αυτά είναι τα βασικά προβλήματα. Και δεν έχουμε αξιολογήσει παρά μόνο με λίγες ad hoc μελέτες ε, των εκ των αντίκτυπο των δραστηριοτήτων έλεγχων της Κομισιόν. Θα ήθελα να σας αναφέρω τώρα κάποια από τα στοιχεία τα οποία αναφέρουμε στην έκθεσή μας για τα δύο έτη που καλύπτει ο έλεγχος, το 2009 και το 2010. Πρώτα απ' όλα να σας πω, στι 19 Ιανουαρίου 2009 εγκρίναμε ένα προσωρινό κοινοτικό πλαίσιο για μέτρα κρατικών ενισχύσεων. Το συνέδριο αξιολόγησε ως περιορισμένη τη χρήση αυτών των μηχανισμών αυτό το προσωρινό πλαίσιο ήταν ε, σε ισχύ μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2011. Για να ανταποκριθούμε στην όλο και μεγαλύτερη ανάγκη εθνικής υποστήριξης στο χρηματοπιστωτικό τομέα, εγκρίναμε ένα ε, καθεστώς ε, κρίσης ό,τι αφορά τις κρατικές ενισχύσεις σε βάση ειδικών ε, καθοδηγήσεων απλουστευμένης επικοινωνίας με τους δικαιούχους και με την συνεργασία μας με εξειδικευμένο προσωπικό στο πλαίσιο μιας ειδικής task force. Καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι η Κομισιόν αντέδρασε έγκαιρα σε ό,τι αφορά τη χρηματοπιστωτική κρίση. Στην Task Force, στην, ε, μάλλον στην έκθεση της Task Force αναφέρονται διάφορες συστάσεις για να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών ελέγχου κρατικών ισχύσεων. Θα πρέπει η Κομισιόν, παραδείγματος χάρη, να είναι πιο προβλεπτική, να υπάρχει μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση ε, για την τήρηση των ε, κανόνων. Θα πρέπει να βελτιώσει η Κομισιόν τις δραστηριότητες παρακολούθησης, να διοργανώσει επίσης δικές της έρευνες με δική της πρωτοβουλία για τις παράνομες εγγυήσεις με ένα πιο συστηματικό και στοχευμένο τρόπο και επίσης θα πρέπει να αυξήσει τη διαφάνεια των διαδικασιών και να επιταχύνει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Θα πρέπει επίσης να δει ίσως η Κομισιόν αν μπορεί να αντλήσει διδάγματα σε σχέση με το πώς χειρίστηκε τη χρηματοπιστωτική κρίση για να βελτιώσει τις συνήθειες μεθόδους μεθόδους και διαδικασίες τη εργασίας. Τέλος, θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη και τις ευχαριστίες μου για την επαγγελματική συνεργασία που είχαμε με τους συναδέλφους και με τους συναδέλφους από την Κομισιόν. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σαντλόβη για την έκθεσή σας. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον εισηγητή, στον κύριο Στάση. Ε, ε, ε, ευχαριστώ Πρόεδρε. Με τη σειρά μου θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την κυρία Σάντοβα και όλη την ομάδα της, την ομάδα της κυρίας Σαντόλοβα. Την ευχαριστώ λοιπόν για την πολύ καλή αυτή παρουσία. Σε μάθα πολλά. η συνεργασία με το Ελεκτικό Συνέδριο είναι πάρα πολύ χρήσιμη εγώ συνήγα κάποια συμπεράσματα, βλέπω ότι υπάρχουν κάποιες συστάσεις. Την περασμένη εβδομάδα επίσης μίλησα επί μακρόν επί την κυρία Σανταλόβα και τον επικεφαλής ομάδας στο Στασβούργο που μου είπαν ότι υπήρχε πράγματι κάποιο μικρό σφάλμα που παρίσφρισε στην πρώτη δική μου σύσταση ε, εγώ θα έλεγα ότι καλωσορίζουμε την ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου και γενικά συμφωνούμε με τις συστάσεις ε, του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Όμως διεξήχθησαν μόνο σε 8 κράτη-μέλη ε, έλεγχοι και αυτό από ό,τι φαίνεται ήταν εσφαλμένο. Πρόθεσή μου ήταν να πω ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο εξέτασε τον τρόπο το γενικότερο με τον οποίο εργάστηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε αυτό το πλαίσιο διενεργήθηκαν οι έλεγχοι σε 8 κράτη-μέλη. Θα αναδιατυπώσω λοιπόν τη σύστασή μου, το σχετικό κείμενο. Στη δεύτερη σύστασή μου λέω ότι είναι πολύ καλό ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντέδρασε γρήγορα και αποτελεσματικά στην οικονομική κρίση και γνωρίζουμε ότι τεράστια ποσά έχουν δαπανηθεί. Η τρίτη σύσταση και ίσως εδώ επικρίνω περισσότερο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υποστηρίζω το ελεκτικό συνέδριο με αυτά που λέω. Λέγω λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να προσαρμοστεί και να η στάση της να είναι πιο ενεργή και νομίζω ότι αναφέρει και το υπογραμμίζει το ελεκτικό συνέδριο αυτό. Επίσης λέω ότι χρειάζονται περισσότερες πληροφορίες που θα χορηγούνται στα κράτη-μέλη και μεγαλύτερη υποστήριξη για τη διάδοση των βελτίστων πρακτικών. Επίσης, τα κράτη-μέλη που δεν είναι πολύ γρήγορα όσον αφορά την κοινοποίηση για τις κρατικές ενισχύσεις πρέπει να πειθαρχηθούν. Χρειάζεται μεγαλύτερη πειθαρχία. Πρέπει να επιβληθεί στα κράτη-μέλη και θα πρέπει να το κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σωστή πει ότι χρειάζεται βοήθεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για κάτι τέτοιο. Και πράγματι υπάρχει ανάγκη για περισσότερου ανθρώπινου πόρου σε αυτόν το τομέα. Αυτό κατάλαβα από την έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου, ότι χρειάζεται προσπάθεια εκεί. Η τέταρτη στασή μου είναι ότι πρέπει να γίνει πιο γρήγορη η δουλειά, να επικρατήσει μεγαλύτερη διαφάνεια και το ελεκτικό συνέδριο το αναφέρει σαφέστατα. Οι διαδικασίε είναι πολύ χρονοβόρες και θα πρέπει να περιοριστούν οι διάφορες ερευνητικές περίοδοι. Έχω ένα ερώτημα προς την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι υπάρχουν κάποια γενικά σχόλια για τα κράτη-μέλη. Θα ήταν δυνατόν να έχουμε μια γενική εικόνα κατά κράτος μέλος σχετικά με το πόσος χρόνος απαιτείται για τα κράτη-μέλη να απεξεργαστούν διάφορα θέματα. Δεν, λέγω δεν ότι χρειάζεται να μας δώσετε τις πληροφορίες αυτές σήμερα, αλλά αν θα μπορούσατε να μας τα δώσετε κάποτε αυτά, να δώσετε αυτές τις πληροφορίες και τη διάρκεια της απαλλαγής ήταν καλό. Πέμπτον, κάτι που ανέφερε η κυρία Σανταλόβα. Συνεχάρη την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι αντιμετώπισε την οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση αποτελεσματικότατα. Ε, μπορούμε να βρούμε κάποια διδάγματα από αυτό. Ε, φαίνεται ότι περισσότερα μπορούν να γίνουν και για τις τράπεζες και για τους απλούς ανθρώπους. Βεβαίως το διακύβευμα ήταν μεγάλο. Αν μπορούν όμως να κινηθούν αποτελεσματικά σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να μάθουμε και τι μπορεί να γίνει και για άλλους τομείς, να αντλήσουμε κάποια διδάγματα. Ερώτηση λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μπορείτε να αντλήσετε κάποια διδάγματα από τον τρόπο με τον οποίο να αντιμετωπίστηκε η οικονομική και η χρηματοπιστωτική κρίση. Να αναπτυχθούν νέες μέθοδοι που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν και αλλού θα μπορούσαμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να έχουμε μια γενική εικόνα ε, και να ενημερωθούμε για οποιαδήποτε νέα μέθοδο. Έκτον, αναφέρομαι στην ανάγκη για μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου για όλους εμπλεκομένους. Δηλαδή ότι αβάσιμες ε, διεκδικήσεις και αξιώσεις πρέπει να αντιμετωπίζονται γρήγορα και θα πρέπει να υπάρξει γενική επιτάχυνση της διαδικασίας εξετάσεως των καταγγελιών και ότι θα πρέπει να διατηρηθούν οι κατάλληλοι πόροι γι' αυτό. μόνο, αναφέρομαι στην ανάγκη για, τους, για περισσότερους ανθρώπινους πόρους και να αντιμετωπιστεί και το θέμα της ε, παρακολούθησης του, χρονικού, του χρονοδιαγράμματος μπορεί να λειτουργήσει για τέλος του έτους ένα σύστημα ενημέρωση διαχείρισης της ε, κοινοποίησης μετά, ε, κρατικέ ενισχύσει είναι πολύ σημαντικές αυτές για τα κράτη-μέλη. Θα πρέπει να βελτιώσουμε την παρακολούθηση ε, των κρατικών ενισχύσεων σαν αφορά το μέγεθο και το πεδίο εφαρμογή. Ε, σύσταση 9. Κάποιο λάθος παρίσφρισε. Ε, η κοινοποίηση και το διαδραστικό λογισμικό, το σχετικό, το ΣΑΝΙ, μεταφράστηκε σε σαρί σε κάποιες γλώσσες. Αντί σανί μεταφράστηκε σαρί, λαθάκι. Ποια είναι η κατάσταση όσον αφορά το σύστημα αυτό, το διαδραστικό, το λογισμικό. Και αν δεν μπορείτε να μας πείτε τώρα, ίσως θα μπορούσατε να μας ενημερώσετε γραπτός κατά τη διάρκεια της διαδικασίας απαλλαγή και θα μπορούσαμε να το λάβουμε υπόψη στην έκθεση του κ. Φιόλνερ για την απαλλαγή. Δέκατη σύσταση. Θα πρέπει να έχουμε μεγαλύτερη αξιολόγηση εκ των υστέρων στον αφορά τις συνέπειες των κρατικών ενισχύσεων και του ελέγχου αυτών επί επιχειρήσεων, αγορών και της ε, οικονομίας εν γέννη προτίθεται να το κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αν ναι, ποιο χρονοδιάγραμμα προβλέπει. Αυτές είναι οι δέκα συστάσεις μου και προτάσεις μου. Ελπίζω ότι μέσω καλής συνεργασίας με το Ελεκτικό Συνέδριο και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ελπίζω ότι τελικά θα προχωρήσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον εισηγητή για όσα μας είπε. Όπως συχνά πρόκειται για ένα μείγμα επένου και επικρίσεων. Υπευλήθη μια σειρά ερωτήσεων προς την Κομισιόν. Θα δώσω το λόγο του Κάτιαν Κρούπμαν από τη Γενική Διεύθυνση Αντανομισμού. Μπορείτε να απαντήσετε τώρα στις ερωτήσεις που σας υποβλήθησαν ή θα μας δώσετε τα αποτελέσματα γραπτά. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κυρία Σανταλόβα, ευχαριστώ κύριε Στάση για την έκθεση, τις δύο εκθέσεις θα έπρεπε να πω και τα διάφορα καλά ερωτήματα και θα ήθελα να καλωσορίσω αυτή την ε, πρωτοβουλία και θα ήθελα σύντομα να δώσω κάποιες απαντήσεις σε όσα έθιξε ο εισηγητής. Καταρχάς, θα ήθελα να πω ότι θεωρούμε εν γέννη ότι η έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου είναι ευπρόσδεκτη και πολλές συστάσεις είναι ορθές, όμως θα ήθελα να πω ευθύ εξ αρχής ότι προφανώς ο έλεγχος κατοικών ισχύσεων σύμφωνα με τη συνθήκη έχει σημαντικό χαρακτηριστικό, δηλαδή υπέχουν ευθύνε και τα κράτη-μέλη δυνάμει τη συνθήκη, ευθύνε και εξουσίε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιορίζονται από τη συνθήκη και νομίζω ότι κάποιο από του τομεί όπου ο εισηγητή σωστά ζητά πρόοδο, αυτοί οι τομεί χαρακτηρίζονται ακριβώ από αυτή τη διάδραση. Δηλαδή, εξουσίε Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπου σκληρέ εξουσίε ε, είναι περιορισμένε και περιορίζονται οι ήπιε εξουσίε από πόρου. Καλό αυτό που υπόθηκε για του πόρου, αλλά στην περίοδο που απετέλεσε αντικείμενο της εκθέσεως του ελέγχου αντιμετωπίσαμε τη χρηματοστική κρίση και έπρεπε να δώσουμε ε, χρήματα για τη μετώπιση της κρίσης. Και κάποια προβλήματα που αναφέρονται στην έκθεση αντικατοπτρίζουν και την εποχή κατά την οποία διεξήφθη έλεγχος. Now, very briefly uh, um, Όσον αφορά τις συστάσεις, καταρχάς, να πω ότι παρόλο που πολλά σημεία της εκθέσεως ήδη μας οδήγησε στο να κινηθούμε, λαμβάνοντας υπόψη σχέδες κανόνες και κανονισμούς, να δώσω κάποια παραδείγματα βάσει και τον ερωτήσεων του κ. Στάες. Πρώτα απ' όλα όσον αφορά τον έλεγχο. Συμφωνούμε ότι πράγματι είναι σημαντικό αυτό. Φέτος διπλασιάσαμε μάλιστα τον όγκο ενισχύσεω που παρακολουθούμε. Θα παρακολουθούμε περίπου το 1 τρίτο όλων των ενισχύσεων που χορηγούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τριπλασιάσαμε και τις, ε, ε τους πόρους που διαθέτουμε. Αυτό έχει συνέπειε. Σα συμφωνούμε απόλυτα ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για την αξιοπιστία του ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων. Δηλαδή ε, θα πρέπει να έχουμε μια πάρα, ένα πολύ καλό στεναρό σύστημα ελέγχου ε, εκ των υστέρων. Ε, μετά τέθη συγκεκριμένο ερώτημα όσον αφορά τη διάθεση των πόρων και πώ μετράται ο χρόνο, ε, ποια συστήματα υπάρχουν, ποιε εφαρμογέ. Ρώτησε και ο Στά, μπορείτε να μα πείτε αν μέχρι το τέλο του έτου αυτό θα, το σύστημα θα λειτουργεί. Έχω την πεποίθηση ότι στο τέλο θα ισχύει το σύστημα που αναφέρατε. Το σύστημα το οποίο αναπτύσσεται είναι το Πέτρα. Ε, ήδη έχει δρομολογηθεί στην αρμόδια Γενική Διεύθυνση. Οπότε θα μπορέσουμε να δούμε πόσο κοστίζει κάθε περίπτωση όσον αφορά του πόρου Έχουμε εισάγει και ένα σύστημα διαχείριση υποθέσεων που μα επιτρέπει να διαθέτουμε όλου του πόρου τη Γενική Διευθύνσεω όσον αφορά τι συγκεκριμένε υποθέσει, συναρτήσει του βάρου αυτών και αυτό οδηγεί σημαντικά κέρδη όσον αφορά την απόδοση τρίτων. Ζητήθηκε να αντιμετωπίσουμε διάφορε καταγγελίε που έχουν συσσωρευτεί και έχουμε μείνει πίσω. Ξεκινήσαμε μεγάλη προσπάθεια πέρσι για να μειώσουμε αυτό, αυτή την υστέρηση που είχε σημειωθεί και έχουμε μειώσει ε, τον αριθμό παλαιών ε, καταγγελιών σημαντικά. Όσον αφορά τη σχέση μας με τα κράτη-μέλη, ζητήθηκε καλύτερη ε, βοήθεια μέσω της διαδόσεως των βελτίστων πρακτικών και να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη που έχουν ασθενέστερα συστήματα. Και εδώ αυξήσαμε τις δραστηριότητε. Εγώ, σαν υποδιευθυντής... Ε, που είμαι υπεύθυνο για τα κράτη-μέλη, έχω επισκεφθεί τα κράτη-μέλη, έχουμε βάλει ε, σημεία επαφή με κάθε κράτο μέλο, είμαστε στενή επαφή με του διάφορου αρμοδίου για την κρατική ενίσχυση στα κράτη-μέλη. Ε, έχουμε προγράμματα κατάρτιση για εθνικού δικαστέ που επίση έχουν ρόλο να παίξουν όσον αφορά τι κρατικέ ενισχύσει και τον έλεγχο αυτών και θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ο κύριο Αλμούνια μάλιστα υπογράμμισε ότι αποτελεσματικό έλεγχο κρατικών ενισχύσεων απαιτεί επίση να παίξουν το ρόλο του για τα κράτη-μέλη. Και στα όρια βεβαίω των πόρων μα θέλουμε να του υποστηρίξουμε, να υποστηρίξουμε τα κράτη-μέλη. Σα δίνω αυτά τα παραδείγματα ως, ε, για να σα δείξω πού έχουμε ήδη προχωρήσει επί τη βάση των ισιών των κανόνων. Και κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό τώρα θέλω να αναφέρω, θα ήθελα να πω λοιπόν ότι πέρα από τη συνθήκη που καθορίζει το βασικό πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύεται από διάφορους κανονισμούς κυρίως το διαδικαστικό κανονισμό που διέπει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζω διάφορε καταγγελίες και ποιε διαδικασίες ε, δρομολογούνται. Νομίζω ότι κάποια από τα ζητήματα που προγραμμίζονται στην έκθεση θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν μόνο πλήρως εάν λάβουμε πολύ σοβαρά, εξετάσουν πολύ σοβαρά τον διαδικαστικό κανονισμό. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν νομίζω ότι είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε και το εξή, ότι απαιτείται από το δικαστικό κανονισμό να ασχοληθούμε με πολύ μικρέ υποθέσει που θεωρείται ότι χρειάζονται ελάχιστο έλεγχο σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ενώσεω, διότι στην πραγματικότητα θα έχουν πάρα πολύ μικρή επίπτωση στην εσωτερική αγορά. Σύμφωνα με του κανόνε, απαιτείται να τι εξετάσουμε τι υποθέσει. Αυτό θα πρέπει να το σκεφτούμε. Παρομοίω, οι παρόντε κανόνε δεν μα επιτρέπουν να ομαδικώ να, να εξαιρέσουμε από έλεγχο κάποιου τομεί στου οποίου παρέχεται ενίσχυση. Ε, και αυτό θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί. Χρειάζεται όμω απόφαση του Συμβουλίου, χρειάζεται αλλαγή ε, του εφαρμοστικού κανονισμού. Αυτό που θέλω να πω λοιπόν είναι ότι είναι πολύ καλά αυτά τα σημεία που αναφέρονται από την έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου και από τον συγητή. Αυτά απαιτούν αλλαγή, αλλαγή του βασικού κανονισμού, των βασικών κανόνων και ω αλμούνια εξέτασε επίσης ε, όλα αυτά τα θέματα υπό το φως του ελέγχου του ελεκτικού συνεδρίου της εκθέσεως του κ. Στάης και αποφάσισε, όπως θα γνωρίζετε από την παρουσίαση του προγράμματος εργασίας το Δεκέμβριο στο Κοινοβούλιο, να ξεκινήσει μεγάλη προσπάθεια εξυγχρονισμού του ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων, όπου όλα αυτά τα ρυθμιστικά θέματα θα μπορέσουν να αντιμετωπιστούν και θα αντιμετωπιστούν θα υποβάλει τις, και θα παρουσιάσει αρχικές ιδέες του στις 2 Φεβρουαρίου σε μεγάλη διάσκεψη που διοργανώνει στις Βρυξέλλες, ακριβώς με θέμα αυτό. Αυτά είναι μηνύματα συγκλίνοντα από την πλευρά μου. Θα ήθελα, αν επιτρέπετε, να υπογραμμίσω κάτι, δύο θέματα μάλλον, όπου εκεί έχουμε αντικειμενικά περιορισμούς. Πρώτα απ' όλα, να γίνει πλήρη εκ των υστέρων αξιολόγηση των οικονομικών συνεπιών κρατικών ενισχύσεων και ελέγχων των κρατικών ενισχύσεων. Είμαι οικονομολόγος επαγγελματίας, θα μου άρεσε πάρα πολύ να κάνω κάτι τέτοιο, αλλά φοβούμαι ότι ο τομέας αυτός των οικονομικών δεν μας επιτρέπει να καθορίσουμε παρκώς ε, ποιες είναι οι συνέπειε για την οικονομία ε, σε όλες τις κατηγορίες συνέπειες των κρατικών ισχύσεων. Αυτό που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα το προωθήσει είναι μια αξιολόγηση των αποτελεσμάτων κρατικών ενισχύσεων και ελέγχων κρατικών ενισχύσεων σε συγκεκριμένου τομεί. Αυτό ήδη είναι, αποτελεί μεγάλη προσπάθεια όμως θεωρούμε ότι είναι κάτι σημαντικό και όπως προανέφερα στα πλαίσια της προσπάθειας εκκριονισμού που ο Αντιπρόεδρος Αλμούνια ανακοίνωσε, Εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να κινηθούμε και ο τρόπο στην είναι ποιον Θα πρέπει να εξετάσουμε ποια είναι η κατάσταση όσο έχει σήμερα. Αυτά λοιπόν. Αυτό είναι ένα όρο που ήθελα να αναφέρω. Περιορισμό δεύτερον. Όσον αφορά τα λεπτομερή στατιστικά στοιχεία, όσον αφορά τη διάρκεια, δεν μπορώ να σα πω σήμερα ότι κατά μέσο όρο, μάλλον πρέπει να πω ότι χρειαζόμαστε πέντε μήνες για να θετηθεί απόφαση βάσει προκαταρκτικής έρευνας ενός μέτρου πριν ξεκινήσει η επίσημη διαδικασία και αν ξεκινήσει η επίσημη διαδικασία αυτό κατά μέσο όρο θα προσθέτει άλλους 21 μήνες. Θεωρούμε αυτό ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά επανερχόμενο σε αυτό που είπα για το διαδικαστικό κανονισμό, αυτή τη στιγμή Αντίθετα από άλλου τομεί πολιτική ανταγωνισμού, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει την εξουσία να ζητήσει πληροφορίε από την αγορά που αφορούν συγκεκριμένε υποθέσει. Δεν μπορεί να ζητήσει κάτι τέτοιο άμεσα από τα κράτη-μέλη ή τα εμπλεκόμενα μέρη. Βασιζόμαστε απόλυτα από τα κράτη-μέλη. Πιστεύουμε το θέμα τη ταχύτητα χρονοδιαγραμμάτων κλπ. Και, και για του πολίτε είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά πρέπει να δούμε ποιοι είναι οι βασικοί κανόνε που διέπουν τι διαδικασίε σε αυτό το πλαίσιο, αν θέλουμε να ε, προχωρήσουμε σημαντικά λεπτομερή στατιστικά στοιχεία από τα κάτι μέλη κατά μία περίοδο που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ασχολείται με τις συνέπειες της κρίσεως σε μία περίπτωση όπου υπήρχαν μεγάλες αποκλήσεις από αυτές που εξετάστηκαν είναι απίθανο να μας οδηγήσει σε γενικά συμπεράσματα. Οπότε καλύτερο θα ήταν να εξετάσουμε τα ομαδοποιημένα στατιστικά στοιχεία και να προσπαθήσουμε μέσω αυτών θα προσπαθήσουμε να διαβιβάσουμε τι πληροφορίε, ε, τι δέουσε, αυτέ που θεωρούμε ότι είναι οι πιο αξιόπιστε κατά τη διάρκεια τη διαδικασία τη απαλλαγή προ τον ε, εισηγητή σα. Ευχαριστώ. Εγώ σα ευχαριστώ κύριε Κόπμαν. Υπάρχουν συμπληρωματικέ ερωτήσει από τα μέλη τη Επιτροπή, από τον εισηγητή, όχι. Σα ευχαριστώ λοιπόν ενκαρδιότατα για τι απαντήσει που μα δώσατε και ελπίζουμε στο σημείο αυτό να μπορέσουμε να προχωρήσουμε γιατί είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό σημείο και μπορούμε να πούμε κάλλιστα ότι ακριβώς η δράση στην κρίση αποδεικνύει ότι μπορεί να υπάρχει ευέλικτη δράση με θετικά οικονομικά αποτελέσματα. Πρέπει να το πει κανένα εδώ εγκομιαστικά, γιατί σε άλλα σημεία χρειαζόμαστε συμπληρωματικές ερωτήσεις ή από κοινού εργασία για να πετύχουμε αυτό που είχαμε. Θα ήθελα από την ευκαιρία να ευχαριστήσω και τη κυρία Σανταλόβα για τη θαυμάσια έκθεσή της. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και διακόπτω τη συνεδρίαση εδώ μέχρι αύριο το πρωί στις 9. Σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ.